Το Πρώτο σημείο στην ημερήσια διαταξή μας. Ψηφοφορία για την ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 106, χορήγηση αδείας για τη χρήση του φθαλικού διεστέρα, DEHP. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για την ένσταση, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Okay, everybody voted. The vote is... Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας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 Okay. Now Εντάξει, να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας της Γενικής Νομοθεσίας για τα Τρόφιμα. Όπως τα ξέρετε, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη γενική αυτή νομοθεσία βάσει τη απόφαση των συντονιστών συστηματικά να προσκαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας ενημερώνει για τη διαδικασία REFIT πριν αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας από την Επιτροπή. Αυτός ο πέμπτος έλεγχος αφορά τον κανονισμό 1972 για τα βασικά πρότυπα και τους στόχους της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Έχουμε τον κύριο Λάντισλαβ Μίκο, Γενικό Διευθυντή της DG Sanko εδώ για το θέμα αυτό και θα του δώσω το λόγο για να μας κάνει την εισήγησή του για τα θέματα αυτά. Και έπειτα θα έχουμε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Καλημέρα σας. Λυπάμαι που χρειάστηκε να με περιμένετε, αλλά ήρθα τρέχοντα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Πάντω δεν είμαι γενικό διευθυντή, είμαι αναπληρωτή γενικό διευθυντή. Ο γενικό διευθυντή μου δεν ήταν σε θέση να έρθει σήμερα. Ευχαριστώ που, μου δώσατε προαγωγή, αλλά ακόμα είναι νωρί. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε επίση την ευκαιρία να κάνουμε μία ενημέρωση για το τι γίνεται με τον έλεγχο αυτό καταλληλότητας της ε, Γενικής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει με τη διαδικασία εξέταση καταλληλότητας ε, στην νομοθεσία πιο ευρέως. Πολύ συχνά μας επικρίνουν γιατί στην νομοθεσία μας αγνοούμε όσους είτε αισθάνονται πως παραβιάζεται η διαδικασία ε, της επικουρικότητας, η αρχή της επικουρικότητας, είτε γιατί η νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη δεόντως ε, τις ανησυχίες και τα δικαιώματα κάποιων ε, πολιτών. Ότι η νομοθεσία μας δηλαδή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τους. Και επειδή η δική μας Επιτροπή θέλει να επιτύχει την καλύτερη νομοθεσία, είπαμε πως θα μπορούμε να παρακολουθούμε την νομοθεσία από την αρχή μέχρι και την εφαρμογή αυτής και να δούμε και πώς επηρεάζει αυτούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των ε, νομοθετικών κειμένων. Είναι μια δικασία στα οποία εμπλέκονται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας τρόπος με τον οποίο επιδιώκουμε την καλύτερη νομοθεσία είναι η εξέταση καταλαλότητας όπου εξετάζουμε κατά πόσο το κανονιστικό πλαίσιο που έχουμε σε κάποιο χώρο είναι κατάλληλο για το χώρο αυτό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ανακαλύψουμε κενά, αντιφάσεις, απαρχαιωμένα μέτρα, υπερχρεωτικές, υπερβολικές επιβαρύνσεις, επικαλύψεις, κτλ. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ μεταξύ του 11 και του 13 ε, κάναμε μια τέτοια εξέταση καταλληλότητας για την αλυσίδα τροφής και τα αποτελέσματα και τα πορίσματα έχουν δημοσιοποιηθεί, μπορείτε να τα διαβάσετε. Βασιζόμενοι σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση, τον Απρίλιο του 2014 ξεκινήσαμε ε, μια διαδικασία εξέταση καταλληλότητας για τον ε, έλεγχο καταλληλότητας γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Είναι το βασικό κανονιστικό ε, πλαίσιο για ολόκληρο το χώρο ε, των τροφίμων, ξεκινώντας από την αρχή της αλυσίδας που είναι η γεωργική παραγωγή και δημιουργεί τα βασικά εργαλεία για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα και για να αντιμετωπίζουμε ε, ε, επίγουσες καταστάσεις μέσω του ΡΑΣΦ ε, και επί τις ιτιστικές κρίσεις όπως και επίσης κρίσεις στο χώρο των ζωοτροφών. Αυτό λοιπόν εξετάζεται και στα κράτη-μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε λοιπόν ε, με μία εξέταση της βάσης, της νομοθετικής και μετά εξετάζουμε τα όσα απορρέουν από αυτή την βάση. Κοιτάμε λοιπόν στον έλεγχο καταλληλότητας αν το πλαίσιο είναι κατάλληλο για να καλύψει το στόχο ολόκληρου του κλάδου τροφίμων και ζωοτροφών εάν ε, όντως συμπίπτει με τις τάσεις στην πολιτική που ακολουθούμε για τα τρόφιμα σήμερα. Η Επιτροπή Γιούγκερ είπε πως θα δώσει προτεραιότητα στον εξυγχρονισμό και στην απλούστευση της τρέχουσας ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος καταλληλότητας γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα εξετάζει τρεις πυλώνες. Το γενικό τμήμα της γενικής νομοθεσίας, δεύτερον τις διατάξεις σχετικά με το ΡΑΦ με τις επίγουσες καταστάσεις και με τη διαχείριση κρίσεων και τις διατάξεις που σχετίζονται με την, με την ΕΣΦΑ. Από τα τρία αυτά σκέλη, μόνο αυτό της υπηρεσίας τροφίμων της ΕΣΦΑ έχει κλείσει, έχει αξιολογηθεί δύο φορές, τελευταία φορά ήταν το 2012. Για να αποκτήσουμε τα πιστήρια που χρειαζόμαστε ε, αναθέσαμε δύο εξωτερικές μελέτες. Πρώτα απ' όλα για το Γενικό Τμήμα της Γενικής Νομοθεσίας και δεύτερον για το ΡΑΣΦ. Όπως επίσης και τις διατάξεις περιχειρισμού ε, ε, έκτατων περιστατικών. Και οι δύο αυτές μελέτες βρίσκονται στη διαδικασία κλεισίματος και θα τις έχουμε αργότερα φέτος για την ΕΣΦΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή ανανεώνουμε την τελευταία έκθεση αξιολόγηση που κάλυψε την περίοδο μέχρι το 2010 σε συνεργασία με την υπηρεσία αυτή, με τα κράτη-μέλη και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε γενικότερη, σε γενικότερο έλεγχο καταλληλότητα, η DG Sante θα λάβει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες όπω επίση και άλλα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα. Ο έλεγχος καταλληλότητα βασίζεται στα πέντε κριτήρια αξιολόγησης. Αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, σχετικότητα, συνέπεια και η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα θα παρουσιαστούν ως έγγραφο εργασίας που θα πάρει την τελική του μορφή το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Για τα συμπεράσματα των δύο εξωτερικών μελετών και για τις ε, αξιολογήσεις της ΕΦΣΑ, όπως αυτές έχουν ενημερωθεί, να σας πω τα εξή. Καταρχήν, σε γενικό επίπεδο η νομοθεσία για τα τρόφιμα έχει πετύχει τους στόχους σας που είναι η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ασφάλεια των τροφίμων έχουν παρατηρηθεί μεγάλες βελτιώσεις σε όλους τους κλάδους εάν συγκριθούν με την κατάσταση πριν ε, έχουμε τη γενική νομοθεσία, δηλαδή η χνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών, η λειτουργία των ε, εμπορευόμενων και συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και για τα ζωοτροφές, όπως επίσης διαφάνεια και εναρμόνιση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη στόχευση των κινδύνων για τα τρόφιμα. Δεν είχαμε συστημικές ε, απώλειες λόγω ε, κάποιων ε, διατάξεων στην νομοθεσία και βέβαια εκεί που υπάρχει χώρος βελτίωσης δεν προκύπτει από τις διατάξεις της νομοθεσίας αλλά σχετίζεται είτε με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και απαιτήσει στη δευτερεύουσα ή δευτερογενή νομοθεσία, στην απορρέουσα νομοθεσία λοιπόν και με την εφαρμογή των υπαρχών των κανόνων από τα κράτη-μέλη. Η αυξημένη παγκοσμιοποίηση και η πολύπλοκη σχέση της προσφοράς του εφοδιασμού και των δικτύων ε, ανεφοδιασμού δημιουργούν θέματα για τα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές και στα πλαίσια αυτά ο βασικός στόχος του ΡΑΣΦ είναι μια γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τούτον τον έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό. Θέλουμε όμω να μειώσουμε τι επικαλύψει και καλύτερη αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ RASF και άλλων δικτύων. Όπω γνωρίζετε, η πρόταση για του επίσημους ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συζητηθεί, μάλλον ξεκίνησε να συζητείται χτες με το Συμβούλιο, έχει αυτό το στόχο κατά νου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κρίση. Αυτό είναι μία από τι προτεραιότητε της νέα Επιτροπής και οι φυστάμενες ε, διατάξεις ε, που ισχύουν και ρυθμίσεις που ισχύουν μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πετύχει της ασφάλειας ε, της υγείας, της ασφάλειας υγείας του καταναλωτή. Χρειάζεται όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συντονισμό αυτής της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές να αυξηθεί. Θα πρέπει η επικοινωνία να αποτελεί τμήμα της διαχείρισης αλλά και της λύσης μιας κρίσης και να μην ε, οδηγεί σε επιβάρυνση μιας κρίσιμης κατάστασης. Το σύστημα γενικά λειτουργεί. Έχουμε κάποιους κλάδους όπου χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή. Καταρχήν, συνέφθα να πούμε ότι χρειάζεται ε, γρηγορότερη ε, παράδοση των αδειών ε, που ε, οι ενδιαφερόμενοι αυτό και για να εξασφαλίσουμε την καινοτομία και γιατί χρειάζεται μια, ένα συγκερασμό τη πραγματογνωμοσύνη που μπορούν να προσφέρουν τα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό, πως θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τους πόρους που σπανίζουν πια στα κράτη-μέλη έτσι ώστε οι εμπειρογνώμονες να είναι σε θέση να συνεργαστούν με την ΕΦΣΑ και ενδεχομένως αυτό να γίνει και στα γραφεία της. Παρόλους τους αυστηρούς κανόνες οι οποίοι συνέχεια επιτηρούνται, πολλές φορές έχει ασκηθεί κριτική στο κατά πόσο είναι απόλυτα ανεξάρτητος ο οργανισμός αυτός, η υπηρεσία αυτή. Να σας πω πως ε, εκεί βρισκόμαστε με τον έλεγχο καταλληλότητας σήμερα. Με χαρά θα ακούσω τη δική σας απόψη και βεβαίως θα απαντήσω και σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσει η συζήτηση, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Σημαντικό βέβαια είναι να πούμε ότι η βελτίωση του τρόπου νομοθέτησης δεν πρέπει να ισοδυναμεί με απορρίθμιση και ότι οι πολίτες μας θέλουν ποιότητα στα προϊόντα τους. Θέλουν να γνωρίζουν την προέλευσή τους, τον τρόπο, ε, τα συστατικά τους, τον τρόπο παρασκευής. Και ταυτόχρονα πρέπει και να προστατεύσουμε τις παραδόσεις μας, τις ε, ονομασίες ε, προέλευσεως και τον τρόπο παραγωγής στις διάφορες περιοχές και τη διαφορά στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πολλές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται συχνά να τηρήσουν τους όρους της. Πολύ συχνά ε, για αυτές γραφειοκρατικής, υπερβολικά γραφειοκρατής νομοθεσίας και δυσκολεύονται να τηρήσουν τις προϋποθέσεις. Είχαμε διάφορα σκάνδαλα, πρώτα απ' όλα το σκάνδαλο με το κρέας. Λόγω είχαμε όλα τα ψυχοδράματα με, τις, ε, με τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, ε, αλλά πέραν του καταναλωτή, ο παραγωγός, ο γεωργός ζητούν πιο λογικές ρυθμίσεις. Πρόσφατα μάλιστα κατέγραψαν οι εφημερίδες, κυρίως στη Γαλλία, μία μελέτη ενώσεων καταναλωτών που αποκαλύπτει πως ε, η σήμανση, οι ετικέτες σε συσκευασμένα προϊόντα ε, προελεύσεως ε, ζωικής, προϊόντα κρέατος, ήταν πολύ ασαφής και μάλλον πηγή σύγχυσης για τον καταναλωτή. Περιμένουμε λοιπόν εμείς ως Κοινοβούλιο ε, να λαμβάνονται υπόψη αυτά που ζητούμε, αυτά που μεταφέρει συχνά και η Επιτροπή για την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν συσκευασμένα προϊόντα κρέατος τα τρανσαμινοξέ επίσης ε, υπάρχει σοβαρό θέμα. Τα έχουν απαγορεύσει οι Ηνωμένε Πολιτείε για λόγους προστασίας από τις καρδιαγκιακές ε, παθήσεις. Θέλω η Επιτροπή να μας πει τι γίνεται με αυτή την υπόσχεση που μας έχει δώσει εδώ και μήνες ότι θα τα απαγορεύσει και εκείνη. Ε, και περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάνιο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω ότι μετά την παρουσίαση αυτή αισθάνομαι ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες μου. Και αυτό γιατί ε, δεν προχωρεί στην υλοποίηση των προσδοκιών του συνόλου των ε, καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη ενημέρωση στο θέμα των τροφίμων, καλύτερη προστασία. Δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής προστασία αυτή τη στιγμή ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε λοιπόν με όλα τα σκάνδαλα και την ε, ανησυχία που όλο και περισσότερο εντείνεται ότι υπάρχει ανάγκη να επιβληθούν ρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε και αυτή ε, την κατάσταση η οποία οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία τους πολίτες. Είπε και η κυρία Γκροστέτ ότι η αλυσίδα των τροφίμων ολόκληρη βρίσκεται σε κατάσταση δυσλειτουργίας, έντονης δυσλειτουργίας, εις βάρος και του παραγωγού και της μικρής εκμετάλλευσης και του ε, εκτροφέα, του κτηνοτρόφου, γιατί σε άλλα σημεία αυτής της αλυσίδας τροφίμων υπάρχουν πανίσχυροι παράγοντες, άνισα πανίσχυροι, οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Άρα χρειάζεται μία σαφής νομοθεσία για την σήμανση και για την ε, ενημέρωση του πολίτη, του καταναλωτή, για το τι είναι δυνατόν να, βρεθεί, να βρίσκεται μέσα στα τρόφιμα που καταναλώνει. Ευχαριστώ. Κυρία Ζούμερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση της κατάστασης. Αντίθετα με το προγραλίσαντα θεωρώ ότι ο καταναλωτής ήδη ε, έχει επαρκή προστασία, ήδη έχει προστασία ε, ως προς τη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια υιοθετούμε και νέα νομοθεσία η οποία ενισχύει αυτή την προστασία. Η ΕΦΣΑ δουλεύει πολύ καλά. Θα υπενθυμίσω το σκάνδαλο με το κρέας από άλογο και το τρόπο και το, ότι διαπιστώσαμε πόσο γρήγορη ήταν η συγκάλυψη της περιεκτικότητας σε κρέας αλόγου των τροφών. Αυτό ήταν το μεγάλο σκάνδαλο. Η δυνατότητα δηλαδή να ε, δηλώνεται ως κάτι άλλο το προϊόν που μπαίνει στην αγορά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι λειτουργεί το σύστημα Υπάρχουν φυσικά περιθώρια και για μεγαλύτερη βελτίωση στα εσωτερικά, ε, στις εσωτερικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ θα πρέπει να δρά πιο γρήγορα και νομίζω ότι αυτό απορρέει και από τα λόγια του εκπροσώπου της Επιτροπής ότι έχει μεγάλη σημασία ο παράγων χρόνος. Φυσικά, εάν έχουμε επαρκές προσωπικό, μπορούμε πιο γρήγορα να επιτελούμε το έργο μας. Και γι' αυτό τίθεται και το ερώτημα. Η ΕΦΣΑ είναι σε θέση να επιτελέσει όλα τα καθήκοντα τα οποία συν χρόνο, της έχουν, ε, έχει επομιστεί με το προσωπικό που έχει στη θέση της. Αυτό πιστεύω πρέπει να το κοιτάξουμε μεγάλη προσοχή γιατί έχει επομιστεί ε, καθήκοντα η ΕΦΣΑ για τα οποία δεν ήταν ε, δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί όπως η παραδείγματι εκστρατεία για ψευδή διαφήμιση σε τρόφιμα ή άλλα ζητήματα Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι ναι, είχε πει η ΕΦΣΑ πως θα προσπαθήσει να τα επομιστεί όλα, αλλά είχε επισημάνει ότι θα έχει ανάγκη σε περισσότερο προσωπικό και αποδεικνύεται αυτό. Πέρασαν χρόνια βέβαια μέχρι να γίνει πρώτη αξιολόγηση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ένας μεγάλος ε, τομέας έχει μείνει εκτός αξιολόγησης και έτσι δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος σε σχέση με την ε, ύπαρξη μιας νομοθεσίας η οποία δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Άλλωστε και η Επιτροπή επαληθεύει το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή ότι έχει υπομειστεί η ΕΦΣΑ το, την επαλήθευση του κανονισμού σε σχέση με τα health claims, δηλαδή με τους ισχυρισμούς περί ε, βελτίωσης ε, της υγείας από τροφές. Πρέπει να κοιτάξει λοιπόν η Επιτροπή. Υπάρχει επαρκέ προσωπικό στη θέση τη ΕΦΣΑ και πώ μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον να τη φορτώνουμε και άλλη δουλειά που δεν είναι σε θέση να επιτελέσει. Κάτι άλλο κύριε Μεγκο, είπατε ότι ο ρόλος της ίδιας Επιτροπής ε, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ως προ τη διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή θεωρείτε με αυτό που λέτε ότι δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες για τη διαχείριση κρίσεων, για ανάληψη δράσης σε διαχείριση κρίσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μήπως θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν και η Επιτροπή περισσότερο προσωπικό. Γιατί τότε θα ρωτούσα δεν αρκεί να ενισχυθεί η ε, επικοινωνία από πλευράς της ΕΦΣΑ, να αναλάβει η ΕΦΣΑ την επικοινωνία σε περίπτωση κρίσεων στο τμήμα της αχύσης κρίσεων. Εκτός και αν κάνω λάθος, θυμάμαι ότι είχε, ασφαλώς βέβαια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλάβει το κομμάτι αυτό το ενημερωτικό, την ε, ενημερωτική εκστρατεία, η ίδια η ΕΦΣΑ και στην υπόθεση του σκανδάλου με το κρέας αλόγου. Ή, εν πάση περιπτώσει, να διατυπώσω αλλιώς την ερώτησή μου, πώς βλέπει έναν ενισχυρημένο ρόλο της ενδεχομένως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ενημέρωση σε περίπτωση κρίσεων. Σε αυτό θα ήθελα κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Και ένα τελευταίο κομμάτι. Γιατί έγινε από ό,τι θυμάμαι δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσίας και ρωτώ εάν αυτή την δημόσια διαβούλευση την έχει αναλύσει το μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακόμα εκκρεμής. Σε αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω να ολοκληρωθεί αυτό το τεστ, αυτή η επαλήθευση αντοχή στο ταχύτερο δυνατό. Έχει κρατήσει πολύ καιρό πια. Εμεί στο Κοινοβούλιο θέλουμε να ανασκοποθούμε και να πιάσουμε δουλειά. Και είναι καλό πλέον ε, στις αρχές του 2016, το πρώτο τρίμηνο του 2016, να καταθέσει προτάσεις η Επιτροπή αλλά εν περιπτώσει τουλάχιστον πριν από τι προσεχείς ευρωεκλογέ. Αυτό το λέω και από την πικρή μα πείρα σε μεγάλα θέματα και το προκείμενο δεν είναι ασήμαντο. Γιατί πάντα το πρόβλημα ήταν ότι δεν προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε τους φακέλους ε, πριν από τις ευρωεκλογέ. Και αυτό βέβαια οδηγούσε σε σοβαρές καθυστερήσεις διότι μετά τι εκλογέ προκύπτει η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου, ένα νέο Κοινοβούλιο δηλαδή, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να επανεξετάσει τι προτάσει και αυτό σημαίνει περισσότερε καθυστερήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χόισλιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ την Επιτροπή που έδωσε τον αρτήριο λάκτισμα στην διαδικασία αυτή. Έχει βέβαια μια, ενέχει μια πολιτική αξιολόγηση. Είχαμε τη συνεργασία με την ΕΦΣΑ την προηγούμενη εβδομάδα Είχαμε την ευκαιρία να τους επισκεφθούμε. Ξέρετε και πολλές φορές μάλιστα, όχι μόνο μία, τους έχουμε επικρίνει. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για τον τρόπο ε, ε, που αναπτύσσει τις εργασίες της Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας, το ΕΦΣΑ, και ε, μας λέει ότι χρειάζεται επιτάχυνση των ε, διαδικασιών συνεργασίας με τους ειδικού. Δεν υπάρχουν επαρκείς εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Δεν διαθέτουν τα κράτη-μέλη τους εμπειρογνώμονες που χρειάζεται η ΕΦΣΑ. Και σε αυτό βέβαια υποφέρει και η ποιότητα της δουλειάς της αλλά και η αξιοπιστία της. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Προκύπτει ως ξεκάθαρο συμπέρασμα των συνομιλιών που είχαμε και βεβαίως τίθεται πάντα το ζήτημα εάν τα καθήκοντα που έχει απομειστεί μπορούν να επιτελεστούν με το υφιστάμενο προσωπικό. Αλλά αυτό είναι και ένα ζήτημα ίσως εσωτερικής διαχείρισης, δηλαδή εάν ικανοποιεί κατά προτεραιότητα τα κύρια καθήκοντά της και στη συνέχεια πηγαίνει στα επιπλέον, στα πρόσθετα. Νομίζω ότι για τα τρόφιμα ε, μπορεί να έχουν μια σειρά από νέα νομοθετήματα στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουν μειωθεί οι ε, νόσοι και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με την ποιότητα τη τροφής που καταναλώνουμε. Άρα ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες αυτές. Γιατί ξέρετε ότι έχει γίνει και η πιο φιλοσοφική συζήτηση για το αν έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές το σκάνδαλο με το κρέα αλόγου νομίζω ότι φώτισε ιδιαίτερα το ζήτημα της διαφάνειας στην αλυσίδα τροφίμων. Για μένα, αντίθετα από ό,τι έλεγε συνάδελφος, δεν αρκεί να ε, διαπιστώνουμε μέσα σε διάστημα τριών ημερών ε, το πρόβλημα και να συζητούμε εάν είναι ζήτημα δηλώσεων ή επιβεβαίωσης από τις αρχές των δηλώσεων. Είχαμε πρόσφατα εδώ στις καντίνες των ευρωπαϊκών οργάνων ζήτημα για το αν το ψάρι που σερβίρανε ήταν αυτό το οποίο αναγραφόταν ή κάποιο άλλο ψάρι ή κάποιες άλλες Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την επαλήθευση της αλυσίδας της τροφής. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί αυτό να σημαίνει κινδύνους που έχουν να κάνουν με κατάλοιπα στα τρόφιμα, κυρίως από ζυζανιοκτώνα, αυτό είναι απαράδεκτο να ανεχόμαστε κατάλοιπα στα τρόφιμα ε, και η παρουσία αυτών ε, στις τροφές μας είναι απόδειξη ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ως προς την αναζήτηση των αιτίων στα προβλήματα. Δεν έχουμε αρκετή συνεργασία με τον κόσμο της γεωργίας, δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Και σε αυτό πρέπει να κάνουμε πιο πολλές προσπάθειες, περισσότερη ενημέρωση, η γεωργική χρήση διζανιοκτώνων αφήνει κατάλοιπα στις τροφές μας, που δεν μειώνονται και νομίζω ότι αντί να το αποδεχόμαστε αυτό σαν κάτι το μοιραίο, πρέπει να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, όταν υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει οι νομοθετικέ διατάξεις να εφαρμόζονται. Και σε αυτό υπάρχει ζήτημα ως προς τα στάση των κρατών μελών. Πρέπει να τα ελέγχουμε πολύ προσεκτικά, πρέπει να ελέγχονται τα κράτη-μέλη ως προς την υλοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας. Και αν χρειάζεται να καλούνται να την βελτιώσουν. Σε αυτό νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εσωτερικά μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση από τις αρχές εποπτείας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πατιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σχολιάσω ένα από τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ζωοτροφών. Η νομοθεσία αναφοράς για αυτές τις ζωοτροφές ορίζει ως επικίνδυνες για την ανθρώπινη κατανάλωση της ζωοτροφές που μπορεί να έχουν ε, επικίνδυνες ουσίες ε, και να προορίζονται ή να περιλαμβάνονται στα συστατικά των ζωοτροφών ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την αντιμικροβολογική αντίσταση. Εδώ λοιπόν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, τα αντιβιωτικά πώς ε, λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη διαδικασία και για σκοπούς προφύλαξης και για σκοπούς ε, αποθεραπείας. Και επίσης για τα ζώα εκτροφής και τα αντιβιωτικά. οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποδεχτεί τη χρήση των αντιβιωτικών αυτών και επίσης την αυξητική ορμόνη και για την καλλιέργεια των γενετικώς τροποποιημένων. Αυτή όμως, ε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει αποδεχτεί όλα αυτά είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Βάσει λοιπόν της γενικής μας νομοθεσία, της διαπραγματεύσεις της TTIP, πώς θα τα πετύχουμε αυτά και πώς θα τα συμβιώσουμε με τα υψηλά πρότυπα για την ε, προστασία της ανθρώπινης υγείας και των ε, συμφερόντων καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων. Ευχαριστούμε κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, το θέμα του ρυθμιστικού πλαισίου αυτού του ελέγχου καταλληλότητας. Η προσπάθεια εναρμόνιση προτείνεται ω προσπάθεια διασφάλιση, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Η πρώτη μου λοιπόν απορία είναι η εξή. Ε, πώς ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι ομοιογενές και τυποποιημένο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις ή κρίσεις ή στοιχεία που έχουν να κάνουν με τοπικά χαρακτηριστικά ή εθνικά, όπως το σύστημα έγκαιρης προποιηδοποίησης όπως προτείνεται το κεφάλαιο 4. Σε περίπτωση κινδύνου ο συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο και με τα κάτι μέλη και τις αρχές τους, τις αρμόδιες αρχές τους είναι απαραίτητος. Όμως το δεύτερο σημείο ε, δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουμε προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή όπως ορίζεται στους γενικούς στόχους ελέγχου ποιότητας προβλέποντας και περισσότερη ευελιξία. Τρίτο σχόλιο και γενική αρχή της ανομοθεσίας η αναδμόνιση με τις διεθνείς συμφωνίες. Εάν θεωρούμε την αρχή αυτή ως αρχή που μπορεί να λειτουργεί σε ένα σύστημα ελεύθερων συναλλαγών και αρκετά διευρυμένου, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται η πιθανότητα να προκύψουν απειλές. Θα πρέπει λοιπόν να μην γίνουμε λιγότερο ελαστικοί και λιγότερο ικανοί να αντιμετωπίσουμε έκτακτες ε, καταστάσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει αυτό υπόψη στην ερμηνεία και τη μεταφορά των διεθνών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Μέλιορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκφράσω τι ευχαριστήσει μου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση τη έκθεση και να ε, κάνω κάποιε παρατηρήσει οι οποίε ε, με ενδιαφέρουν για περαιτέρω ε, πληροφορίες. Είχαμε με μια μικρή ομάδα που ήταν και ο πρόεδρος μέλος να, ε, την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους εκπροσώπους της ΕΦΣΑ και τον νέο πρόεδρο κύριο Ούλο για να, και να διαπιστώσουμε ότι ιδιαίτερα ενδιαφέρεται να δώσει απαντήσεις και να αποκρούσει κατηγορίες οι οποίες ε, εξ αρχής είχαν εκφραστεί ότι εκφράζει τα συμφέροντα της ε, βιομηχανίας, ότι παίζει με σημαδεμένα η τράπουλα κτλ. Και είδαμε την προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων με επιστημονικές γνώσεις που θα έπρεπε να διαθέσουν τα κράτη-μέλη χάρη στην οποία θα, μπορούσαν, θα μπορούσε να αναβαθμίσει και την αξιοπιστία της η ΕΦΣΑ. Άρα χρειάζεται τους εμπειρογνώμονες η ΕΦΣΑ και θα ήθελα να ρωτήσω εσείς πώς μπορείτε να την υποστηρίξετε στην ε, προσπάθειά της αυτή για να ενισχύσει την εικόνα της και την αξιοπιστία της. Και μια άλλη ερώτηση, έχουμε ένα γενικό δίκαιο για την ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υλοποίηση όμως, ε, η αντιμετώπιση του από τα κράτη-μέλη και υπάρχουν δυνατότητες με την επικουρικότητα να γίνουν ε, επιμέρους επιλογές σε κάποια σημεία, είναι ε, διαφορετική. Η υλοποίηση είναι διαφορετική ή θα έλεγα λίγο συγκρίσιμη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω έχετε τελικά σαν στόχο μια πιο ενιαία εφαρμογή για την ενιαία προστασία της δημόσιας υγείας του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά για να έχει όλο και καλύτερη ποιότητα ζωής ο καταναλωτής και να μειώνεται στο δυνατόν η παρουσία των λεγόμενων πολιτιστικής φύσεως ε, ε, νόσων τι κάνετε λοιπόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου αυτό το ενιαίο κατά τα άλλα δίκαιο να εφαρμόζεται και κατά τρόπον ενιαίο για να εξασφαλίζονται τα ίδια δικαιώματα για όλους τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now Miss Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω σε ένα σημείο. Ψηφίσαμε μια έκθεση το Φεβρουάριο φέτος για την προέλευση των ε, συσκευασμένων κρεάτων. Νομίζω πως ε, εκτός από το θέμα της ασφάλειας, ε, της υγείας των καταναλωτών, χρειάζεται και πραγματική διαφάνεια για την επιλογή που αγοράζει ο καταναλωτής κάποιο τρόφιμο. Νομίζω ότι τους οφείλουμε αυτή τη διαφάνεια για να γνωρίζουν τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν. Περιμένω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο σημείο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους να ζητούν το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να απαντήσει. Να σας ευχαριστήσω για μια εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων με ιδιαίτερη ένταση η οποία αναφέρεται σε πολλά από τα στοιχεία που μας απασχολούν. Είναι πλούσια και όμορφη συζήτηση που γίνεται για τη Γενική Νομοθεσία, για τον ε, Γενικό Νόμο για τα Τρόφιμα όχι μόνο για τα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε τι που άκουσα. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν πως υπάρχει εξή τάση και είναι γενικότερη, δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υπάρχει μια τάση να προσπαθούμε να εισάγουμε νέα νομοθεσία για να το αντιμετωπίσουμε. Παράλληλα, πολλοί λένε πως η Ευρώπη έχει υπερβολικά πολλή νομοθεσία. Αφενός λοιπόν πιέζουμε για νέα νομοθεσία και αφετέρου ε, προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των νομοθετικών κειμένων. Η μόνη λύση είναι πρώτα καταρχήν να εξετάσουμε το τρέχον νομικό πλαίσιο. Καταρχήν καλύπτει ή όχι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, εάν το καλύπτει, το καλύπτει επαρκώς με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η βασική αρχή της ε, προσπάθειας που κάνουμε με τον έλεγχο καταλληλότητας. Όταν μιλάμε για έλεγχο καταλληλότητας γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, και σας υπενθυμίζω κάτι που όλοι γνωρίζετε, είναι μιλάμε για μια πυραμίδα νόμων, πάνω από χίλιες εφαρμοστικές πράξεις, κατεξουσιοδότηση πράξεις, νομοθετικά κείμενα που βασίζονται στις αρχές που έχουμε θεσπίσει στην Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα. Κοιτάμε λοιπόν τη βάση. Η βάση είναι εντάξει, οι αρχές που διέπουν τη βάση αυτή είναι σωστές, είναι σωστά ε, τα όσα χτίσαμε σε επίπεδο θεσμών και μετά θα ανέβουμε την πυραμίδα προς όλη την υπόλοιπη ε, απορρέουσα νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε και εκεί πολλά από τα όσα θίξατε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και θα μπω και στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνατε, πως πολλά έχουν αντιμετωπιστεί ήδη σε ένα πακέτο το οποίο προτάθηκε πριν από μερικά χρόνια και το οποίο συζητάμε ακόμα. Μιλήσατε και εσείς, τη συζήτηση, ε, μιλήσατε και εσείς για τους επισήμους ελέγχους, για τους επίσημους ελέγχους, ε, όπου ακόμα η συζήτηση δεν έχει κλείσει και δεν έχουμε εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομερή συζήτηση κάθε μίας νομοθετικής πράξης και μεμονωμένων θεμάτων, γιατί αυτό ξεπερνά το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου καταλληλότητας, ε, μιλώντας για συγκεκριμένη λύση, συγκεκριμένο πρόβλημα. Ενώ η ερώτηση εδώ είναι οι αρχές οι οποίες διέπουν τη γενική νομοθεσία επαρκούν, λειτουργούν σωστά ή χρειάζεται να αλλάξουν έτσι ώστε όλη η υπόλοιπη νομοθεσία να έχει μια στέρεη βάση. Να απαντήσω όμως και σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, που κατέγραψα κατά τη συζήτηση. Για τα λιπαρά, ναι, είναι πρόβλημα. Θα τα δείτε στην έκθεσή μας και θα τα συζητήσουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Το Δεκέμβριο νομίζω θα κληθούμε να το απαντήσουμε. για την οθεία. Όντως η οθεία στα τρόφιμα είναι πρόβλημα, αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί με έναν ακόμα κανονισμό. Η νοθεία είναι εξορισμού μία απάτη εκτός νόμου. Άρα λοιπόν περισσότεροι κανόνες δεν θα μας βοηθήσουν, εργαλεία χρειαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε ε, τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουμε αυτές τις ε, πρακτικές και να τις καταστήλουμε. Τι δεν είχαμε στο παρελθόν. Διάφορα στοιχεία κομβικά τα οποία προτείνουμε στον ε, κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους και νομίζω ότι υπάρχει γενικότερη στήριξη από πλευράς Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν πως μόλις κλείσει η συζήτηση εκεί θα αποκτήσουμε τα εργαλεία για την πάταξη της νοθείας κάνετε πολλά σχόλια για την ΕΦΣΑ. Θα το απαντήσω όλα μαζί. Καταρχήν τα σχόλια που λένε πως η ΕΦΣΑ αντιμετωπίζει πάνω από 500 αξιολογήσεις το χρόνο με προσωπικό 500 περίπου υπαλλήλων και 10 ε, επιστημονικές ε, επιτροπές, εγώ πρέπει να σας πω πως τα πάνε καλά. Παρόλες επικρίσεις για τη διαφάνεια και τα λοιπά και τα πραγματικά προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε, δεν έχετε άδικο. Όμως, κατά τη γνώμη μας η νομική βάση είναι επαρκής. Επαρκεί το, το προσωπικό. Ναι. Η αξιολόγηση που κάναμε απέδειξε πως το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον αριθμό προσωπικού και υπαλλήλων, αλλά από τα εξή. Ένα, το αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή χρειαζόμαστε τους κορυφαίους επιστήμονες της επιστημονικές επιτροπές της ΕΦΣΑ και παράλληλα, και παράλληλα με συγχωρείτε, αυτοί πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Μα ξέρετε πως οι επιστήμονες εργάζονται κυρίως σε project τα οποία χρηματοδοτούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πώς είναι δυνατόν να είσαι κορυφαίος επιστήμονας και μέσα στα 10 χρόνια, τα πιο πρόσφατα 10 χρόνια, μην καμία επαφή με τις επιχειρήσεις του κλάδου. Διαφορετικά θεωρούνται ως ενδεχομένως ευάλωτες επιέσεις. Τελικά έχουμε ή πολύ νέους επιστήμονες ή επιστήμονες ταξιούχους γιατί αυτοί οι οποίοι είναι δραστήριοι και κορυφαίοι που έκαναν ένα-δύο project με την τάδε εταιρεία τα τελευταία χρόνια αποκλείονται γιατί δεν θέλουν να εξωστραγιστούν από τα μίνδια ως λομπίστες των ε, επιχειρηματικών ε, συμφερόντων. Χρειάζεται λοιπόν η συνδρομή των κρατών μελών στο σημείο αυτό. Κάτι που δεν ανέφερε είναι επίσης πως η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να πάει σε έναν επιστήμονα και να πει «εσένα θέλω». Όχι. Πρέπει να επιλέξουν από αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πως οι οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται είναι οι κατάλληλε έτσι ώστε να έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή επιλογής υποψηφίων στην ΕΦΣΑ. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα νομικής βάσης. Η νομική βάση είναι εντάξει. Είναι η, είναι η πρακτική εφαρμογή, η δεξαμενή επιστημόνων και η πίεση στο να έχουμε ε, ε, να μην έχουμε επιμόλυνση από τους εταιρικούς κύκλους. Αυτά μας δυσκολεύουν. Και στο πλαίσιο αυτό νομίζω πως η ΕΦΣΑ κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως όλοι μπορούμε να βελτιωθούμε. Αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Για τις αιτήσει. Για τα θέματα βοτανικής, ε, για τον βοτάνικα, με συγχωρείτε, ε, δεν είναι πρόβλημα ελλείψης τελέχωσης της ΕΦΣΑ. Εκεί έχουμε μία σύγκρουση δύο νομοθεσιών. Οπότε, αν εφαρμόσουμε τους ε, υφισταμένους κανόνες χωρίς να εξετάσουμε τις επιπτώσεις, θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Δηλαδή, θα τα έχουμε βάλει όλα το ίδιο κουτί χωρίς να επιτρέψουμε σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αιτήσεων, ποια είναι σχετική, ποια όχι. Αν όλα τελικά τα αρνηθούμε, τι κάναμε. Να δούμε λοιπόν την ουσία εδώ και το περιεχόμενο και όχι να πούμε πως δεν έχουμε τη δυνατότητα ή τις ε, δυνάμεις. Όχι, πρέπει απλώς να βρούμε τον τρόπο, τη σωστή προσέγγιση. Και εδώ είμαστε εκτός πεδίου γενικής νομοθεσίας. Είναι σε άλλο επίπεδο που θα πρέπει να βρεθεί η λύση. Εσωτερικές διαδικασίες χρήζουν βελτίωση στην ΕΦΣΑ, ναι. Το είδαμε και με το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου και εμείς συμμετέχουμε. Όπως και με την διοίκηση της ΕΦΣΑ, πρέπει να σας πω πως στην οργάνωση της ε, δουλειά τη γίνονται πολλές αλλαγές. Το είπε και ο εκτελεστικός, εκτελεστικός διευθυντής πρόσφατα. Οπότε νομίζω πως αυτές οι βελτιώσεις θα γίνουν. Για το ρόλο που παίζει σε μια κρίση η ΕΦΣΑ, να σας υπενθυμίσω, τι κάναμε και τι ψηφίσατε εσείς. Που είναι σωστό. Αποφύσαμε στην Ευρώπη να χωρίσουμε την αξιολόγηση κινδύνου από την διαχείριση κινδύνου. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση. Η ΕΦΣΑ έχει ρόλο να παίξει στην αξιολόγηση του προβλήματος, αλλά δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει τμήμα της διαχείρισης του προβλήματος. Αυτός ο ρόλος έχει ανατεθεί από την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και στις αρμόδιες αρχές αυτών. Και θα πρέπει έτσι να συνεχίσει. Να χρησιμοποιήσουμε την επιστημονική, ε, το επιστημονικό δυναμικό της ΕΦΣΑ για να μας συμβουλεύει, αλλά μέχρι εκεί. Όχι σε επίπεδο διαχειριστικό λοιπόν. Καμιά φορά έχουμε μια επικάλυψη σε στιγμές κρίσης. Αυτό είναι φυσιολογικό, κατανοητό. Γιατί δεν χρειάζεται καν μέρες στη διαθέσεις σου για να αποφασίσεις τι θα κάνεις, ώρες μόνο. Αλλά προσπαθούμε αυτή τη διάκριση να τη σεβόμαστε σε κάθε στιγμή. Τώρα, Γενική Νομοθεσία Τροφίμων. Έλεγχος καταλληλότητας. Ένα έχει καταλήξει κάποια συμπεράσματα, επαναλαμβάνω. Όχι ακόμα, αλλά πρώτο τρίμηνο του 2016. Ναι, πρώτο τρίμηνο του 2016 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα σας παρουσιάσουμε τα σχετικά συμπεράσματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Τώρα λάβαμε τις μελέτες τις οποίες αναθέσαμε για να συλλέξουμε πληροφορίες και αξιολογούμε το ποια θα είναι η περαιτέρω δράση μας. Νομίζω ότι μέσα στους επόμενους δύο-τρεις μήνες θα έχουμε ένα σχέδιο κειμένου και μετά θα περάσει εσωτερική διαβούλευση κτλ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 λοιπόν θα σας παραδώσουμε το κείμενο αυτό. Um, yeah, uh, I think it was also several times... Νομίζω αρκετές φορές <clears throat> αναφέρθηκε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Ενώ το νομοθετικό πλαίσιο ε, είναι επαρκές, μπορεί να το πει κανείς αυτό, σε μερικέ ε, περιοχέ, σε μερικού τομεί υπάρχει δραματική κατάσταση ω προ την υλοποίηση. Και στην Ευρώπη το θέμα είναι ότι η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου ανατίθεται στι εθνικέ αρχέ των κρατών μελών. Ενώ η ευρωπαϊκή σκοπιά, το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ένα ρόλο ελέγχου. Πρέπει να είμαστε τελείω σαφεί ω προ αυτό. Να θυμίσω λοιπόν ω προ την επιβολή και την υλοποίηση έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο ονομάζεται ε, γραφείο ε, επισυντηστικό και εκτινατρικών θεμάτων, ε, το οποίο συνδράμε τις Εθνικές Αρχές των Κατών Μελών στην υλοποίηση των επιμέρους κανόνων για την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί αναλύουμε και αποτιμούμε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Ευρωπαϊκής ε, Νομοθεσίας, δίνοντας απόκριση στα κράτη-μέλη όπου χρειάζεται και όπου μας ρωτούν για το τι πρέπει να γίνει για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι απαντήσεις είναι κάποιες φορές λιγότερο ή περισσότερο καλές, αλλά συνήθως επιτυγχάνουμε κάποιο αποτέλεσμα και ε, υπάρχει αρκετά καλά συντονισμένη συνεργασία του ευρωπαϊκού επίπεδου με τις εθνικές αρχές το ερώτημα για το αν οι κανόνες που προβλέπονται από την νομοθεσία μας που έχουν πολύ ψηλά πρότυπα ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων και πόσο αυτοί μπορούν να συμφιλειωθούν με τις διαπραγματεύσεις μας για το TTIP. Δεν θέλω να ανοίξω πάλι μια συζήτηση που έχουμε κάνει επανειλημμένως, αλλά είναι αλήθεια και το έχουμε ξαναπεί. Ο ρόλος της συμφωνίας TTIP δεν είναι να αποδυναμώσει το δικό μας επίπεδο ασφάλειας ο στόχο είναι να βρούμε ακριβώ το σημείο ισορροπία, το χώρο που μπορούμε να έχουμε το επίπεδο ακόμα και αν καταλήγουμε σε αυτό μέσω διαφορετικών μεθόδων. Επίση, να δούμε κατά πόσο στο μέλλον υπάρχει περιθώριο, χωρί να ε, υποβαθμίσουμε τα πρότυπά μα, να συγκλίνουμε με του Αμερικανού, ώστε να υπάρξουν εισαγωγέ και εξαγωγέ από του μεν προ του δε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν υπήρξε ουδέποτε θέμα, ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν είπα κάτι τέτοιο, ότι θα ξανασυζητήσουμε τα όρια της Ευρώπης λόγω των διαπραγματεύσεων TTIP. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό και συμμετέχω προσωπικό στις διαπραγματεύσεις, οπότε μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Για, τις, ε, για τους κινδύνους της ε, αντίστασης, το θέμα αυτό δεν το καλύπτει ακριβώ η Γενική Νομοθεσία. Δεν αυτό αυτό λοιπόν ένα από τα αντικείμενα των ελέγχων καταλληλότητα. Υπάρχουν όμω αρχέ που ε, προτείνονται από τη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα, οπότε αυτό θα το αντιμετωπίσουμε, θα το ε, εξετάσουμε στα πλαίσια των συζητήσεων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που μπορεί να περιλαμβάνουν συστατικά από φάρμακα η σχετική πρόταση θα ολοκληρωθεί το 2016 και θα προβλέψουμε και ένα πρόγραμμα δράση, το δεύτερο μέρο του προγράμματο δράση για την ερχόμενη χρονική περίοδο. Αξιοποιώντα και τι αρμοδιότητέ μα που μπορούν να προκύπτουν και για τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τι ζωοτροφίε, την ομοθεσία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση δηλαδή. Ε, μετά οι ερωτήσει για την εναρμόνιση και την ευθυγράμμισή μας με διεθνείς κανόνες. Πολύ σημαντική ερώτηση και έχει δύο πτυχές. Πρέπει να σας θυμίσω και πάλι ότι από τη μια είμαστε υποχρεωμένοι βάσει των κανόνων να τους εφαρμόζουμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά Στη δέσμη μέτρων για τους κτηνιατρικούς και τους επίσημους ελέγχους δεν ήταν απόλυτα σαφές. Προσπαθήσαμε να, να περιλάβουμε στην ομοθεσία μας όλε μα τι σχετικέ υποχρεώσει, οπότε συμμορφούμαστε πλήρω τελικά με τι διεθνεί συμφωνίε. Υπάρχει όμω και μια άλλη σημαντική πτυχή. Ω πρωταγωνιστέ ε, στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών παγκοσμίω, θα πρέπει να είμαστε και επιτυχημένοι στην μετάφραση ε, και την μεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων που είναι πολύ αυστηροί προς τις διεθνείς συμφωνίες. Δηλαδή το δικό μας επίπεδο ασφαλείας να το ε, με τα λαμπαδέψουμε και στις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες φορές για τους Ευρωπαίους πολίτες οι διεθνείς κανόνες είναι λιγότερο αυστηροί από ό,τι αυτοί που θέλουμε να ε, ισχύουν για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε και του διεθνεί κανόνε να καλύψουμε με τη δική μα την νομοθεσία, αλλά από την άλλη είναι προ όφελο των ευρωπαϊκών κανόνων. Είναι αυτοί που ε, καθορίζουν τα πρότυπα για του υπόλοιπου ε, συμμετέχοντε τη διεθνή διαπραγματεύσει. Αυτά ε, ήταν τα στοιχεία με τα οποία ήθελα να απαντήσω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Πρόεδρο, εμείς... Σα ευχαριστώ και εγώ <clears throat> για τη λεπτομερή απάντηση. Μπορούμε πιστεύω πια να περάσουμε στο επόμενο. Θα μας αναμερίσει στη διάταξη που είναι ανακοίνωση καινοτομία και τεχνολογικών εξελίξεων στην γεωργία, στην εκμετάλλευση, στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο κύριος Τσόλφολη είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη της Πέθρου, που είναι καθήλυνα αρμόδια, έχει προβλέψει μια έκθεση πρωτοβουλίας που στόχο έχει, αντικείμενο μάλλον έχει, την προώθηση της ε, καινοτομίας το ε, στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντο. Ζητάτε λοιπόν ε, μια δική μα γνωμοδότηση που αντιμετωπίζει βασικά ζητήματα για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μα είναι πώ θα θρέψουμε τον πλανήτη. Ένα θέμα που αφορά και τη διεθνή, είναι αντικείμενο και τη διεθνού έκθεση του Μιλάνου φέτο. Ε, και όπου έχουν προταθεί διάφορες λύσεις. Ένα θέμα λοιπόν, μια γενική αρχή την οποία θέλω να παραλάβω και έχουμε λάβει ως σημείο για την έκθεση είναι ότι ο ρόλος του Γιώργου είναι να παράγει πρόθυμα αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει ε, να ε, προστατεύεται και η γονιμότητα του εδάφους ε, για σκοπούς γεωργικούς και όχι για, περιτούς, για χρήσεις του εδάφους να υποβαθμίζεται η ποιότητα αυτού. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι προκλήσει έχουμε μπροστά μα να αντιμετωπίσουμε. Αυξήνεται ο πληθυσμό του πλανήτη που θα φτάσει τα 9,6 δι ε, ανθρώπους μέχρι το 2050 με την ε, κατά συνέπεια αύξηση της ζήτησης σε τρόφιμα παγκοσμίω. Η απόκριση στην ζήτηση αυτή θα πρέπει να ε, μας οδηγήσει στην επισητιστική ασφάλεια την εξασφάλιση επαρκούς και υγιούς ποσότητας τροφίμων. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε και του πολύτιμου πόρου του πλανήτη για τι ερχόμενε γενιέ. Θα πρέπει λοιπόν επί τη ουσία να παράγουμε περισσότερο, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Με λιγότερη χρήση νερού, ενέργεια, λιπασμάτων, ζυζανιοκτώνων και φυτοφαρμάκων. Ένα νέο λοιπόν γεωργικό μοντέλο αυτό τη κυκλική οικονομία ε, είναι μια εναλλακτική που πρέπει να την ε, λάβουμε υπόψη πλέον η γη χρειάζεται 1,5 χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις της μετά από την καλλιέργεια ενός χρόνου. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τα απόβλητα τροφίμων που ε, μας οδηγούν στον... Ε, πετάμε ε, ένα εκατομμύριο τρακόσες χιλιάδες τόνους ε, τρόφιμα επισίως ενώ 800 εκατομμύρια βρίσκονται σε συνθήκες πείνας και λιμού, καθώς και υπάρχει και πρόβλημα υπέρβαρου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παχυσαρκίας. Θα πρέπει λοιπόν τα απόπλητα τροφίμων να δορίζονται αντί να πετώνται, ε, αντί να αποκομίζονται σε ειδικέ φιλανθρωπικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν την ε, νέα τους διανομή. Και θα πρέπει να δούμε και ποια είναι αυτά τα υποπροϊόντα της γεωργίας που μπορούν να, να αξιοποιήσουν την ε, ύπαρξή τους για σκοπούς παραγωγής ενέργειας λόγου χάρη και για χρήσεις διακριτές από αυτές της απλής αποκομιβής. Θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με την βιώσιμη παραγωγή και καλλιέργεια για να έχουμε επαρκή παραγωγή και επισητιστική ασφάλεια, την απαραίτητη δηλαδή ποσότητα τροφίμων, να έχουμε προστασία της ανθρώπινης υγείας και την απαραίτητα ποιότητα των τροφίμων. Αλλά να προστατεύουμε και την υγεία των ζώων με, προστα... με σεβασμό του περιβάλλοντος, αποφυγή της απώλειας της βιοπικιλότητας, την αποφυγή της εκπομπής ε, ρήπων ε, για την ατμόσφαιρα και βεβαίως όλα αυτά, αυτόν τον υψηλό στόχο, μπορούμε να το πετύχουμε με την καλλιέργεια της καινοτομία και της έρευνας, ε, δίνοντας έμφαση στους νέους. Με μια νέα οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερα εισοδήματα από την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και με διαφανείς συνθήκες στην αγορά, με ε, σαφή ετικετοθεσία και αναφορά της χώρας προέλευσης. Πρέπει να στηρίζουμε τους γεωργούς στην πράξη, με μια γεωργία εξυγχρονισμένη, καινοτόμο, που να είναι και βιώσιμη, να είναι εφή, smart και να είναι βιολογική, να είναι επίσης ακριβίας, να βασίζεται σε, ε, στη χρήση υπολογιστών και ρομποτικής. Αυτά τα στοιχεία για τη νέα γεωργία είναι σημαντικά για την ανανέωση, την γενεαλογική των ε, γεωργών της μερίδας αυτής του πληθυσμού και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γύρασης του πληθυσμού στις περιοχές της Πέτρου, την ε, απερίμωση και τις ορεινές περιοχές που εγκαταλείπονται εκεί μπορεί να δημιουργηθούν πραγματικοί κίνδυνοι για την υδροπολογική ισορροπία το... της επικράτειας ε, των ε, κρατών μελών και του εδάφους τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες γεωργικές πρακτικές, να επιδιώξουμε τη διάδοσή τους και ακόμη και τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμετελεύσεις που είναι η πλειονότητα στην Ευρώπη να τις στηρίξουμε πολλές φορές δεν βρίσκονται στην ε, σωστή, στο σωστό κύκλο δικτύωσης για την καινοτομία. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, ε, αξιοποιήσουμε τις, να εφαρμόσουμε μάλλον αρδευτικές και γεωργικές πρακτικές που να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε και τις κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά για να αποφύγουμε και τις μεταναστευτικές ροές εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον κλιματικούς πρόσφυγες. Εδώ λοιπόν στάθηκα απλώς στα βασικά σημεία της έκθεσης για την καινοτομία στην Γεωργία. Μπορούμε βεβαίως να βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόταση με τις απαραίτητες τροπολογίες οι οποίες πρέπει να υποβληθούν ως τις 27 Νοεμβρίου. Είμαι βέβαιος ότι θα ε, προσφέρετε κι εσείς τις δικές σας απόψεις και τοποθετήσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Κέρστιγκερ. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Λαμπία, αντικαθιστώ την σκιώδη μας, την κυρία Πέτια σήμερα, μια και δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Έχω τις γραπτές της παρατηρήσεις και θα σας τις μεταφέρω. Θέλει να υπογραμμίσει ένα-δύο σημεία που χρειάζονται χρειάζεται να αναδειχθούν περισσότερο, να ενθαρρύνουμε δηλαδή την καινοτομία και κυρίως την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και τις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους γεωργούς. Πιστεύει επίσης ότι πρέπει να υποστηριχθεί η καινοτομία, κυρίως εκείνη η οποία τίνει στη μείωση του κόστους παραγωγής με την περιφερειοποίηση του κόστους της κατανάλωσης ενέργειας, υδάτων και άλλων πρώτων υλών ή με την ενσωμάτωση στη ροή της κυκλικής οικονομίας. Πιστεύει επίσης ότι η καινοτομία θα πρέπει να συμβάλλει σε πιο αηφόρο ε, παραγωγή τροφίμων με την παραγωγή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη και την διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Η υπερβολική παραγωγή τροφίμων και η συσσόρευση τροφίμων στις αγορές είναι μια λαθασμένη επιλογή όπως μας λέει η σκιώδη συγγήτρια και λέει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν πιο καινοτόμα μοντέλα στον τομέα της γεωργίας για την προστασία των καταναλωτών και της ποιότητας της γεωργικής υγείας ως σημαντικού πόρου. Εάν αυτό το παραγνωρίσουμε, εκτιθέμεθα στον κίνδυνο και να μην δώσουμε λύσεις και να καταδικάσουμε την γεωργική μας παραγωγή για το μέλλον. Χρειαζόμαστε αηφορία στις πολιτικές και τις δράσεις μας και για το καλό των μελλοντικών γενναιών. Θα ήθελα λοιπόν η σκιωδησηγήτρια να παρακαλέσει την εισηγητή να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Νίκολσον, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του πολύ σωστά υπογραμμίζει την μεγαλύτερη ουσιαστικά πρόκληση που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέα στην Ευρώπη, την ασφάλεια των τροφίμων. Η παραγωγή τροφίμων θα χρειαστεί να διπλασιαστεί έως το 2050 για να ικανοποιεί την ζήτηση που θα έχει ε, φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα με αυτό. αλλά αυτό με τους ίδιους πόρους. Έτσι λοιπόν αν εντατικοποιήσουμε την παραγωγή των τροφίμων με αηφορία μπορούμε ή μάλλον για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε και τεχνολογία και επιστήμη ε, ως βάση των αποφάσεων που θα λάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κοιτάξουμε ιδιαίτερα τις τεχνικές ε, παραγωγής ακριβίας, precision farming και δεδομένα ε, επιστημονικά για την καθοδήγηση αυτής. Οι παραγωγοί θα έχουν νομίζω να ρόλο να διαδραματίσουν ασφαλώς, θα, θα χρειαστεί να καταρτήσουν και να εκπαιδεύσουν τους νεότερους γεωργούς, να τους εξοικειώσουν και με τις ε, νέες βέβαια τεχνολογίες και η ενίσχυση της κοινοτομία δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην απόκτηση της τελευταίας ε, τεχνολογικής δυνατότητας Έχουμε πολλές ομάδες ε, τεχνολογίας, 160 τον αριθμό στη δική μου την εκλογική περιφέρεια που μελετούν τις εφαρμογές τεχνολογίας στη γεωργία και μπορούν να επιτρέψουν και ε, με την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιση των πρακτικών μεταξύ των γεωργών. Η καινοτομία λοιπόν για τις ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως έχει και η διαχείριση, το management για την ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων, κάτι το οποίο σημαίνει ουσιαστικά διαφύλαξη, συντήρηση και του πιο ικανού αποδοτικά ε, αλλά πρέπει να επεκταθεί και στην προστασία του πιο αδύναμου ε, σε απόδοση σαφές για το BBC, κυρίε και κύριοι, ιδιαίτερα μια, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπομπή για τα αποφάγια, για τα απόβλητα τροφίμων. Η... Ε, το βασικό μήνυμα της εκπομπής αυτής ήταν ε, αντί να πετάμε τα τρόφιμα, τα αποφάγια μας ή να τα βάζουμε στον σκουπιδοφάγο, να τα ξαναχρησιμοποιούμε για να παράγουμε νέα τρόφιμα. Πρέπει αυτό το κομμάτι να το ε, κοιτάξουμε μεγάλη προσοχή για να μπορέσουμε να διασώσουμε την παραγωγή τροφίμων μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την ε, τόσο καλή συνεισφορά του. Νομίζω σωστά δίνει έμφαση στα βασικά σημεία που θα πρέπει να σταθούμε ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μιλώ και εκ μέρου τη κοιόδου συγκεντριά μα, τη κυρία Τόραβλετ, που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, ίσω να υπερβαίνουμε κάπω τα όρια ω προ την ομοδότηση τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, όμω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι ριζοσπαστικά να αλλάξουμε την κοινή αγροτική πολιτική τελικώ αντί απλώ να ε, προβλέψουμε ένα σύστημα στηρίγματος των εισοδημάτων των γεωργών. Ένα σύστημα που επιτρέπει στους γεωργούς να προχωρήσουν στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ίσως να εκτεβαίνουμε κάπως τα όρια. Όμως η καινοτομία είναι ένας από τους τομείς κλειδιά για να διασφαλίσουμε επαρκή παραγωγή τροφίμων για το μέλλον. Εφόσον θα φτάσουμε σχεδόν τα 10 δις ε, Ανθρώπου στον πλανήτη. Καινοτομία βέβαια δεν σημαίνει αναγκαστικά νέε πρακτικές πάντοτε. Πρέπει να είμαστε και λίγο πρακτικοί στην ε, σκέψη μας. να δείξουμε ότι έχουμε πρακτικό μυαλό. Εάν αναζητούμε καινοτόμου τρόπου για την ε, γεωργία και τι καλλιεργίε, ήδη θα έχουμε τεράστια κέρδη ω προ την παραγωγικότητα τη Ευρώπη. Η ανταλλαγή των ε, καλοπρακτικών είναι ήδη λοιπόν κάτι σημαντικό θα ήταν μια καινοτόμω προσέγγιση. Ένα άλλο τομέα, και αυτό είναι στην καρδιά των ενδιαφερόντων τη Επιτροπή τη δική μα, είναι να βεβαιωθούμε ότι αυξάνεται η παραγωγή χωρί να διακινδυνεύει το περιβάλλον. Εάν δούμε αυτό που συζητήσαμε και χθε στην έκθεση Nature δηλαδή για το περιβάλλον και τους, ε, τα οικοσυστήματα και του οικοτόπου, θα δούμε ότι η εντατική γεωργία είναι μια από τι βασικέ αιτίε απώλεια βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια σαφή πρόκληση μπροστά μα. Από τη μια θέλουμε περισσότερη παραγωγή και από την άλλη πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτή την απώλεια βιοποικιλότητα. Όμω σίγουρα οι καινοτόμε τεχνικέ στη Γεωργία και απαραίτητε είναι, αλλά και η καλύτερη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπω ήδη υπάρχουν. Ίσως απλώς να χρειάζεται να ε, απεντατικοποιήσουμε τις πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ, θα ε, υποβάλω τις σχετικές τροπολογίες για αυτή την τόσο ήδη ισχυρή έκθεση στην τοποθετησή σας. Ευχαριστούμε ο κ. Χόισλιν. Ναι. Θα εύχομαι και εγώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα στα οποία τοποθετείται. Είχε και πέρσι το θέμα αυτό η Επιτροπή Γεωργίας και παρακολούθησα την επιχειρηματολογία εκεί γιατί και έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί και στην Επιτροπή Γεωργίας θεωρούν ότι τεχνολογία ισοδυναμεί με φυτογίνα προϊόντα, με χρήση νέων λοιπασμάτων και το καθεξής. Θεωρούν ότι αυτό είναι η πρόοδος και είναι λάθος προσέγγιση γιατί η δυτικοποίηση δεν πρόκειται να μας πάει μακριά. Πιστεύω λοιπόν και το έθιξαν κάποιοι συναδελφοί ότι αυτό το είδος της γεωργίας έχει σημαντικές παρενέργειες, απώλεια βιοπικιλότητας και ε, απεμπλουτισμό των εδαφών. Έχουμε μέχρι τώρα με μεγάλη ανεμελιά διαχειριστεί τους σπόρους μας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για το μέλλον έτσι. Για μένα καινοτομία γεωργική, γεωργία στραμμένη στο μέλλον σημαίνει ένα νέο γεωργικό μοντέλο με λιγότερο input, με καλύτερη διαχείριση και με διασφάλιση. Που είναι ικανή να διασφαλίσει δηλαδή την ασφάλεια των τροφίμων. Εάν λέτε ότι θα χρειαστεί να αυξήσουμε την παραγωγή τροφίμων κατά 70% όπως ακούστηκε τώρα, αυτό θα απαντούσα ε, προϋποθέτει ότι θα συνεχίσουμε την κατανάλωση και τα, τα μοντέλα κατανάλωση που έχουμε εμείς τώρα. Και δεν νομίζω ότι πρέπει δεν είναι δυνατόν ολόκληρο ο κόσμο να τρέφεται με τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν οι, Αμερικα... οι Ευρωπαίοι, ακόμα και χειρότερα οι Αμερικανοί που έχουν μεγαλύτερη ακόμη ε, κατανάλωση κρέατος και να θεωρούμε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα είναι βιώσιμο. Η κατανάλωση γάλακτο, κρέατος που έχει η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε επίπεδο παγκόσμιο, γιατί τελευταία δεν κάνει και σε κανέναν καλό. Είναι τέτοια τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης ε, πρωτεΐνης και τελευταία ανάλυση ζωικής πρωτεΐνης και τελευταία ανάλυση αυτό δεν εξυπηρετεί κανέναν γιατί με, το, με τη μαζική παραγωγή οι τιμές όλο και πέφτουν. Άρα λοιπόν τα μοντέλα κατανάλωσης θα πρέπει να είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Στις χώρες μας πολλά είναι τα ε, τρόφιμα τα οποία πετάμε στα σκουπίδια. Σε άλλες ε, οι... οι συνθήκες είναι τέτοιες γιατί δεν υπάρχει ασφαλής αλυσίδα ψήξης και γίνεται η εκαθάριση των προϊόντων τροφίμων σε πολύ ε, νωρίτερο επίπεδο και έτσι δεν φτάνουν καν ορισμένα παραπροϊόντα τροφίμων μέχρι τον καταναλωτή. Επίσης πρέπει να κοιτάξουμε το ζήτημα της γνώσης που πάει χαμένη, της παράδοσης και των ε, προϊόντων, του, του, των γνώσεων, των πολιτιστικών που χάνονται με τη γύρανση του γεωργικού πληθυσμού και την απώλεια αυτών. Ευχαριστώ κύριο Μπάλτσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. το σχέδιο γνωμοδότησης είναι πολύ σαφές για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Κάποιες από τις προκλήσεις αυτές ε, αντιφάσκουν μεταξύ τους βεβαίως και ο συντάκτης της νομοδότησης ε, σημείωσε την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, κάτι που θα σημάνει ανάγκη περισσότερης παραγωγής τροφίμων. Στην Ευρώπη πάντως προσπαθούμε να παράγουμε τρόφιμα ποιότητας. Να μην ε, λησμονούμε ότι μνήα υπάρχει στην, στο σχέδιο νομοδότησης ότι μια άλλη λειτουργία που πρέπει να λάβει η Γεωργία είναι να διατηρήσει την Ήπεθρο, τον πληθυσμό της. Αυτό δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βρούμε λύσεις για την απερίμωση της Ήπεθρου, ε, για την ε, φυγή από τη, τα χωριά και τις μικρές πόλεις της επαρχίας. Θα πρέπει Επίσης, να δούμε και τις τεχνικές που αναφέρθηκαν και τη χρήση της ρομποτικής. Εξ όσων γνωρίζω, η ρομποτική χρησιμοποιείται στη γεωργία για να παραχθούν γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα και όλος ιδιαίτερος ε, φύτρες σόγιας. να δούμε τι συμβαίνει με εκμεταλλεύσει όπου όλη την καλλιέργεια την φέρνουν εις πέρας μηχανήματα. Τι θα γίνει όμως ε, στην περίπτωση αυτή εάν το δούμε σε συνάρτηση με το άλλο θέμα, την απερίμωση το, της υπαίθρου. Δεν βρίσκω λοιπόν ότι αυτό ε, συμβαδίζει με τους στόχους μας, ίσως πάντως να μην κατάλαβα πολύ καλά το σχόλιο του εισηγητή. Ευχαριστούμε κυρία Πύρικ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα χτε τα όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας γιατί συζητούσαμε ένα παρόμοιο, παρόμοιο θέμα. Μιλούσαμε για την ΚΑΠ του μέλλοντος και πρέπει να σας πω πως ο αγροδιατροφικός τομέας είναι μεγάλος στην Ευρώπη και παρόλα αυτά δεν εμπλέκονται καθόλου στη συζήτηση του θέματος. Χθες με τον εκπρόσωπο της ΕΤΕ μιλήσαμε για την ε, συμφωνία για το κλίμα και είπαμε 30% βιώσιμη ενέργεια. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για θέματα όπως τα λιπάσματα, για την αποθήκευση αυτών, για τα ε, αζωτούχα, ε, για τα θέματα της οδηγίας για το καθαρό νερό, για τον ατμοσφαιρική, την ατμοσφαιρική ρήπανση του αέρα. Θα ήθελα λοιπόν να μην προσπαθούμε για 20 χρόνια να προσθέσουμε κάτι τέτοιο στη συζήτηση. Θέλουμε καινοτόμα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τους παραγωγούς και επίση για καινοτόμα μέτρα, να μιλήσουμε για καινοτόμα μέτρα στον αγροδιατροφικό τομέα για να καλύψουμε και μια σειρά άλλα ζητημάτων που θα πρέπει να βρεθούν συνοδηγία αυτή. Υπάρχουν συνοδηγία για τα λοιπάσματα όπω επίση και για τα απόβλητα αλλά μην ξεχνάτε πω έχουμε μικρέ εκμεταλλεύσει, τι οποίε με κάποιο τρόπο θα πρέπει να στηρίξουμε και να το κάνουμε και σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συγητή και να επισημάνω την ολόψυχη υποστήριξή μου προς την έκθεση. που αποτελεί μια ευκαιρία να ενισχυθεί η καινοτομία και να βελτιωθεί η εικόνα του γεωργικού τομέα. Κάτι για το οποίο συζητήσαμε και χθε στην Επιτροπή Γεωργίας, όπου εκφράστηκαν φόβοι για την ε, απασχόληση ε, της θέσης εργασίας, ε, το όριο πρασινίσματος και ούτω καθεξής. Πρέπει όμως να δώσουμε μια ευκαιρία να προχωρήσει αυτή η υπόθεση γιατί ο κλάδος της γεωργίας θεωρείται ως ένας πεπαλαιωμένος, μη αποτελεσματικός ρηπογόνος, ζημιογόνος για τις κλιματικές συνθήκες τομέας. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Και πρέπει να βελτιωθούν βέβαια κάποια πράγματα, αλλά και αυτή είναι η φιλοδοξία που θα πρέπει να καλωσορίσουμε θερμά, ε, της εκθέσεως για το πρασίνισμα, για την αξιοποίηση των για τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας και για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της εικόνας ολόκληρου του γεωργικού τομέα, στον οποίο αφιερώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μέσα από τον μεγενθετικό φακό της γεωργίας βλέπει ο πολίτης το, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε τις κατευθύνσεις ώστε να την βλέπει πια σαν κάτι το καινοτόμο, σαν κάτι που, σε ένα τομέα που βελτιώνει και δεν επιδεινώνει την κατάσταση, δεν πετάει σκουπίδια, ε, στα σκουπίδια τα τρόφιμα που παράγει πλεονασματικά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον εισηγητή και όλους όσοι συνεργάζονται. Ευχαριστώ κύριε Τουλαχάγεφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, ε, να σας πω λοιπόν πως για τα σημεία τα οποία αναφέρατε, ναι, έχουμε τρισεκατομμύρια εκατομμύρια τόνους τρόφιμο που πετάμε στα σκουπίδια. Ναι, θα πρέπει αυτό να εμφανίζεται κάπου, ε, κάπου ξεκάθαρα, δηλαδή ποια είναι η σπατάλη τροφίμων και το είχα πει και στον επίτροφο Χόγκαν ότι θα πρέπει αυτό κάπου να φαίνεται. Πριν όμως προωθήσουμε νέα μέτρα, θα πρέπει να επαληθεύσουμε το κατά πόσο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή τα θέματα του, του πρασινίσματος, του greening στην ΚΑΠ. Γιατί καλό είναι να προωθούμε την βιολογική γεωργία, αλλά δεν είναι η μοναδική που υπάρχει σήμερα και καλό θα ήταν να προωθήσουμε παράλληλα και την ε, γεωργία η οποία σέβεται πολύ το περιβάλλον. Για το σημείο 8, αυτό ήταν το σημείο 6, θέλω να κάνω μια παρατήρηση για την καινοτομία, να σας πω πως η πρόσβαση στο ίντερνετ, στις ε, ζώνες της ε, υπαίθρου, είναι ένας δείκτης προόδου έτσι ώστε η Γεωργία να σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και θα πρέπει αυτό το big data, τα μεταδεδομένα δηλαδή ως έννοια να μπουν ε, και στον χώρο της Γεωργίας. Ε, Βεβαίω πάντα με την απαραίτητη τήρηση του απορρίτου. Ευχαριστούμε. Τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρο και όδη συγκεντρία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόφολη για την γνωμοδότησή του και επειδή ανακεφαλαίωσε πολλά από τα σημαντικά σημεία που αφορούν την Γεωργία. Ε, εδώ συμμεριζόμαστε πολλές από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον για να προσαρμοστεί η γεωργία στις κλιματικές αλλαγές και να καλύψουμε τις ανάγκες της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Νομίζω πρέπει να τάξουμε την ευκαιρία για να προβλέψουμε και άλλες αρχές στην αναμοδότηση αυτή που μπορούν να κατευθύνουν καλύτερα τις μελλοντικέ μας δράσεις. Αναφέρθηκε από κάποιου συναδέλφου ο ρόλο τη βιοπικιλότητα, η προστασία τη βιοπικιλότητα ε, και ε, αναφέρεται βεβαίω το έγγραφο του εισηγητή. Όμω δεδομένων των ε, ορίων, χαρακτήρων για τη σύνταξη τη γνωμοδότηση, θα μπορούσε να δοθεί και περισσότερο χώρο στο τελικό κείμενο, στην τελική εκδοχή του κειμένου, σε αυτή την τόσο σημαντική διάσταση, την προστασία τη βιοπικιλότητα δηλαδή, να την ελαχιστοποιήσουμε έστω την απώλειά της ή και να την ε, ανατρέψουμε πλήρως. Αναφέρθηκε επίσης προηγουμένως το θέμα της ε, αποδυνάμωσης του εδάφους. Θεωρώ ότι ως Ευρωπαίοι και όπως ε, ανέφερε και στην αντίστοιχη εκθεσή του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος, ο Περιβάλλοντος, θα πρέπει να δούμε το θέμα της ε, αποδυνάμωσης των ε, εδαφών. Επίσης, οι τεχνολογικές λύσεις όπως η ο μεριακός εμπλουτισμός κάποιων ειδών ή η αντίσταση, η μικροβολική αντίσταση κάποιων ειδών μαζί με την ε, παραγωγή ζωοτροφών και την απεξάρτησή μας από τις εισαγωγές, από τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά δεν αρκούν το επίπεδο της παραγωγής. Ε, θα παρέμβουμε βέβαια, αλλά πρέπει να παρέμβουμε και σε επίπεδο κατανάλωση ώστε στις αγορές να προωθούνται τα τοπικά προϊόντα, κάτι που είναι σκόπιμο και λογικό και για τους γεωργούς, ώστε να μπορούν να επενδύσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά και να πάψει και εντατική καλλιέργεια. Επίσης να βρούμε τις κατάλληλες ε, τεχνολογικές λύσεις για να προάγουμε την βιολογική γεωργία και να έχουμε και μια επιπλέον περιβαλλοντική προσέγγιση ώστε να διαδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα και ζωικά είδη και να προστατευτούν ταυτόχρονα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε και τώρα λόγο ε, στην Επιτροπή, στον κύριο Πίτερ, για, να, για να ακούσουμε και τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Κύριε Πίτερ, δεν είστε εδώ. Όχι. Η Επιτροπή απουσιάζει. να αφήσουμε την δυνατότητα στον εισηγητή μας, τον κύριο Τζόφολη, να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι πραγματικά συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Θα δούμε πώς μπορούμε να τις περιλάβουμε τις διαφορετικές απόψεις, ε, βελτιώνοντας την πρόταση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το μέλλον, δεν πρέπει να φοβόμαστε την κοινοτομία και την έρευνα. Στοιχεία καθοριστικά και για τη γεωργία μας, αλλά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τι ερευνητικέ μας προσπάθειες και τα πορίσματά τους να τα κατευθύνουμε στη νέα θεώρηση για την ανάπτυξη που όλοι να πτήσουμε ε, και όλοι μαζί οραματιζόμαστε για την Ευρώπη και για την ε, παγκόσμια κοινότητα. Πέραν της κρίσης που διανύουμε τώρα, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και κρίση αξιών, προοπτικών και ιδεών, Όλα αυτά μας προσκαλούν και μας υποχρεώνουν να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 29 ε, Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα καλέσω τον κύριο Μπερτολίνη επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο της ε, Έρμες να έρθει εδώ στο Προεδρείο και θα συζητήσουμε την γνωμοδότηση της ΙΑΚ για την πιθανή καρκενογένεση από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργαμισμένων προϊόντων κρέατος κάτι που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Για το λόγο αυτό θα του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο του, το λόγο για να μας παρουσιάσει τα πορίσματα της ε, μελέτης αυτές και να έχουμε συζήτηση μεταξύ μας. Κύριε Μπερτολίνη. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή ΕΝΒΗ του Ευρωκοινοβούλιο για την πρόσκλησή του που μας επιτρέπεται λοιπόν να παρουσιάσουμε καλύτερα τα πορίσματα της μελέτης μας, ε, της, ε, του οργανισμού μας πριν από λίγες εβδομάδες για τα θέματα του καρκίνου. Ε, είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα τις τελευταίες εβδομάδες με πολλά άρθρα και πάρα πολλές ε, τοποθετήσεις, απόψεις και σχόλια από διαφορετικές σκοπιές και φορείς. Να σας πω λίγα περισσότερα για τις μονογραφίες της IARC και τι εννοούμε. Μιλάμε για ένα είδους εγκυκλοπαίδειας για τα διάφορα είδη καρκίνου και τις καρκινογόνους παράγοντες ε, και ερευνούμε ουσιαστικά τι προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους και τι όχι. Ε, δεν πρόκειται για μια απλή αξιολόγηση ναι ή όχι. Ε, υπήρξαν πολλές αξιολογήσεις με την έκθεση, την περιβαλλοντική, την εργασιακή, την, τους χημικούς σωματικούς και βιολογικούς παράγοντες, όλα αυτά αποτιμήθηκαν από κοινού και 118 παράγοντες ταξινομήθηκαν ως καρκινογόνοι με την απάντηση ναι ή όχι καταρχάς και μετά 360, 360 εντοπίστηκαν ως ενδυνάμει καρκινογόνοι παράγοντες. Βάσει των στοιχείων αυτών η Εθνική Αρχή και οι διεθνείς φορεί μπορούν να αντιδράσουν λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα η αποτίμηση, η αξιολόγηση της, ε, για το κόκκινο κρέας και τα επεξεργασμένα προϊόντα προέκυψαν λόγω της σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΡΚ, η οποία αποφάσισε ποια θέματα πρέπει να εξετάσει. Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία δίνει συστάσεις για ουσίες και ε, στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν. Υπήρξαν αρκετέ επιστημονικέ μελέτε τι τελευταίε δεκαετίε για το συγκεκριμένο ζήτημα και οι τελευταίε συστάσεις από τον ΠΟΗ του 2002 ήταν ήδη ξεπερασμένε και περάσει καιρό. 22 λοιπόν ανεξάρτητοι επιστήμονε, ε, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να υπογράψουν μια κοινή δήλωση για να αντικατασταθούν εφόσον υπήρξε, υπήρχε παραμικρή σύγκρουση συμφερόντων, ε, εξέτασαν πάνω από 800 μελέτες επιδημιολογικές, ε, ζωικές και από ε, πειράματα in vitro. Αυτό κράτησε έξι μήνες και τα αποτελέσματα συντάχθηκαν και κλεισμέναν των θυρών ε, επί σειρά εβδομάδων. Τώρα, ποια είδη προϊόντων εξετάσαμε από μια κόκκινο κρέας, δηλαδή βόλιο, χοιρινό, μοσχαρίσιο και αλόγου, ε, αρνή, ε, κατσίκι, ε, αλλά όχι άγρια θυράματα ή πουλερικά. Δεν υπήρχαν αρκετέ μελέτε για την περίπτωση, για τι τελευταίε περιπτώσει. Έπειτα τα επεξεργασμένα προϊόντα αναλύθηκαν και αυτά. Οποιοδήποτε προϊόν κρέατο, κάποιε φορέ και με πουλερικά τα οποία αναμειγνύονται στη, στα στατικά των προϊόντων. Επίση με την τεχνική τη του καπνίσματος, της ε, προσθήκης ε, μπαχαρικών και ούτω καθεξής της πάστοσης και ε, ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν είδαμε ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στους ανθρώπους βάσει των στοιχείων που έχουμε εντοπίσει και κυρίως καρκίνο του ορθού. Ε, εδώ επίσης για το κόκκινο κρέας είδαμε ότι είναι ενδυνάμει ίσως κατά πάσα πιθανότητα καρκινογόνο για τους ανθρώπους αν και δεν έχουμε αρκετά αποδεκτικά στοιχεία ούτε όμως μπορούμε και να αποκλείσουμε κάποια από τα πελέσματα των ε, μελετών και των πειραμάτων. Υπάρχουν ε, διαφορετικά μεθοδολογικά ζητήματα, διαφορετικές προϋποθέσεις σε κάποιες από τις μελέτες οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο. Και ο σχετικός κίνδυνος ώστε κάποιος να παρουσιάσει καρκίνο του ορθού ε, καταναλώνοντας προϊόντα επεξεργασμένου κρέοντος είναι 18%. Είναι η αναλογία αυτού που καταναλώνει και αυτού που δεν καταναλώνει για κάθε ημερήσια κατανάλωση 50 γραμμαρίων ε, προϊόντων επεξεργασμένων ε, από κρέας. 18% λοιπόν τις 100 πιθανότητες να παρουσιάσει καρκινό Ε, να πω λίγα λόγια και για τον ορισμό τι ε, συμφωνήσαμε και τι αποφασίσαμε και τι ε, μεταδώσαμε και στον τύπο. Έχουμε μια ομάδα προϊόντων που παρουσιάζουν πολλές, ε, πολλούς καρκινογόνους παράγοντος. με την αρχική ερώτηση ναι ή όχι αν η ουσίες ή τα συντοτικά αυτά είναι καρκινογόνα. Και μιλάμε για το γενικό πληθυσμό και τις περιπτώσεις να παρουσιαστεί καρκίνο στο γενικό πληθυσμό, σε απόλυτους αριθμούς. Μιλάμε για έναν ορισμό που θέτει στο ίδιο επίπεδο το κόκκινο κρέας ή κάποια άλλα ε, προϊόντα. Όπως το κάπνισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάπνισμα ή το αλκοόλ ή η ατμοσφαιρική ρήπανση έχουν την, ε, τις ίδιες συνέπειες για την υγεία όπως ε, το κόκκινο κρέας ή τα επεξεργασμένα προϊόντα. Βλέπετε εδώ τις διάφορες υποκατηγορίες που μελέτησε η Γιάγκελκ ε, η πρώτη είναι εκεί που υπάρχει βεβαιότητα ότι προκαλείται καρκίνο. Η δεύτερη είναι ότι είναι εκεί που υπάρχουν κάποιε ε, μεγάλε πιθανότητε. Έπειτα μερικέ πιθανότητε, έπειτα λιγότερε και τέλο καμία πιθανότητα. Εάν τα συγκρίνουμε όλα αυτά μεταξύ του, καταλήγουμε ότι ο κίνδυνο για τον πληθυσμό ω προ τι ουσίε, την ίδια κατηγοριοποίηση, τη πρώτη δηλαδή ομάδα, βλέπουμε για τα επεξεργασμένα προϊόντα αύξηση των πιθανότητων παρουσίαση καρκίνου του ορθού κατά 100%. Ενώ η κατανάλωση 20-30 τσιγάρων ημερησίω αυξάνουν την πιθανότητα παρουσίαση καρκίνου των πνευμόνων κατά 20-25 φορές. Δηλαδή 200 2.500%. Ε, Επίση το ίδιο για την κατανάλωση 4-5 ποτηριών κρασιού μπύρα ημερησίω που θα μπορούσε να αυξήσει τον καρκίνο του φάρικα κατά 180%. Ε, εδώ λοιπόν, αν δούμε του απόλυτου αριθμού από μελέτε για τον γενικό πληθυσμό, βλέπουμε από το σύνολο 8 εκατομμυρίων κρουσμάτων θανάτου από καρκίνο παγκοσμίω, 1 εκατομμύριο φροντιστών ε, ε, στο κάπνισμα, 600.000 στο αλκοόλ, 400.000 στην ατμοσφαιρική ρήπανση, 50.000 μάλλον στο κοκκινό κρέα, και λέω μάλλον γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρω, και 34.000 στα επεξεργασμένα προϊόντα. Βλέπετε λοιπόν πόσε ε, είναι οι πιθανότητε. Α δούμε μια συγκεκριμένη χώρα ω παράδειγμα και Μπορώ να σα το εξηγήσω και με περισσότερε λεπτομέρειε αν χρειαστεί. Αν δούμε το Ηνωμένο Βασίλειο λόγου χάρη και υποθέσουμε ότι, ο καθένας, ότι όλοι έπαβαν το κάπνισμα από τη μια μέρα στην άλλη, θα είχαμε 64.500 λιγότερε περιπτώσει θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων. Καρκίνο που δεν εμφανίζεται καθόλου. Εάν όλοι έπαβαν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος υπερκαζεμένων προϊόντων, θα είχαμε 8.800 λιγότερα κρούσματα. Θα με ρωτήσετε λοιπόν γιατί συγκρίνουμε τις 64.500 έως, προς τις 8.800 περιπτώσεις αυτό γιατί δεν καπνίζουν τόσοι όσο οι άνθρωποι που καταναλώνουν κόκκινο κρέα σε επεξεργασμένα προϊόντα. Είναι λοιπόν μικρότερο αριθμό των περιπτώσεων, αλλά ισχύει για τον ευρύτερο πληθυσμό. Οι αριθμοί μπορεί να είναι κάπω παραπλανητικοί από αυτή την έννοια, αλλά σα δίνουν μια ε, εικόνα τη τόξεων μεγέθου. Γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά. Ε, γιατί το κόκκινο κρέα μπορεί να είναι καρκινογόνο. Πρώτα απ' όλα α δούμε την χημική διάσταση. Το κρέα, περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μόριο το οποίο ονομάζεται ε, αίμα, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο είδος σιδήρου και μπορεί να ε, μιμηθεί τα μόρια των εντέρων. Αυτό να ερεθίσει τα μόρια των εντέρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ε, μικρών όγκων και τελικά μακροπρόθεσμα στη δημιουργία καρκίνου. Υπάρχει λοιπόν καρκινογόνος παράγοντας. Το ίδιο Το ίδιο για κάποια ζωτούχα συστατικά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, ε, κάποιες συγκεκριμένες χημικές ουσίες, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο και η παρασκευή των τροφίμων, η υψηλή θερμοκρασία λόγου χάρη, εάν ψήνουμε το κρέας υψηλή φωτιά, μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως πολυκυκλική, αρωματική ή υδρογονάτρακες. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι είπε και ο τύπος τα τελευταία τις τελευταίες ημέρες με τα δημοσιεύματά του. Είπαν ότι δεν είναι κάτι, κάτι τόσο καινούργιο, το ξέραμε και λίγο, το υποψιαζόμασταν. Ναι, υπήρχε υποψία ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα θα μπορούσαν να είναι ενδυνάμικα κοινογόνα. Αυτό αυτό ήταν λίγο πολύ γνωστό σε κάποιε χώρε, αλλά υπήρξαν και χώρε που πήραν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Κάποιε λίγε χώρε, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προτείνει να μην καταναλώνεται ιδιαίτερα ε, μεγάλη ποσότητα επεξεργασμένων προϊόντων. Η Σουηδία προτείνει συγκεκριμένη ποσότητα για την κατανάλωση κόκκινου κρέατο ανά εβδομάδα. Η Ολλανδία σκοπεύει να περιορίσει τα επεξεργασμένα προϊόντα και η Αυστραλία επιτρέπει μόνο την κατανάλωσή του κάποιε φορέ και σε μικρέ ποσότητε. Όμω η τελευταία μελέτη από το 2003 λέει ότι όσοι δεν είναι φυτοφάγοι ε, καλούνται να μετριάσουν την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατο λουκανικών, ε, σαλαμιού, μπέικον ε, και χειρομεριού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα μα προσχολήσει και πάλι. Για να ολοκληρώσω, η αποτίμηση, η αξιολόγηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη στι συστάσει για μια υγιή διατροφή. Το κρέα είναι πηγή και για πρωτενε και για σίδηρο και για βιταμίνε και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Αυτό ε, το τονίζουμε στη μελέτη μα, δίνοντα και τι απαραίτητε πληροφορίε. Γενικώ η σύστασή μα σε αυτό το χρονικό σημείο για μια υγιή διατροφή είναι να αποφεύγουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατο, διότι είναι καρκινογόνα και επί περιλαμβάνουν υψηλό επίπεδο θερμίδων που μπορεί επίση να δημιουργήσει άλλα προβλήματα όπω ε, την παθησαρκία και ούτω καθεξής. Να περιορίζεται καταναλώση κόκκινο κρέατο, να φροντίζουμε άλλε πηγέ να μα παρέχουν την να καλύπτουν τι ημερήσει ανάγκε μα σε πρωτενε, σίδηρο και βιταμίνε, να τρώμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και να περιορίσουμε την κατανάλωση αλατιού και ζάχαρης καθώς και να αποφεύγουμε το αλκοόλ. Έτσι έχει κατάσταση σήμερα και περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τα σχόλια και τι παρατηρήσει σα. Σα Σας ευχαριστώ πολύ <clears throat> για την παρουσίασή σα. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Με την κυρία Καπεσόν Ρουίς που ζήτησε το λόγο. Gracias, presidente. Bueno, Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας προφανώς η διατροφική ασφάλεια είναι αποφασιστική αποφασιστική για την υγεία μας και θα πρέπει να αναφέρεται πάντα το στοιχείο αυτό. Όμως θα ξεκινήσω με μία επίκριση γιατί χωρίς να μπω στην ουσία του συμπεράσματος της μελέτης πρέπει να πω πως Νομίζω ότι ήταν απερίσκεπτος ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιήθηκε το πόρισμα αυτό. Γιατί όπως είπατε κι εσείς θα έπρεπε να έχετε κλείσει με το γεγονός πως μια ισορροπημένη διατροφή είναι η καλύτερη λύση με μια σειρά από τρόφιμα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται. Το να λέτε πως ε, Όντως η υπερβολική κατανάλωση μεταποιημένων τροφίμων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του παχαίου εντερού. Εντάξει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε το συμπέρασμα αυτό, όταν δεν έχουμε καν πρόσβαση στις μελέτες οι οποίες ε, χρησιμοποιήθηκαν, δεν ήταν σωστή. Γιατί το συμπέρασμα είναι το πιο σημαντικό. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει λεχθεί διαφορετικά. Και επί ουσίας δεν έχω τα επιστημονικά δεδομένα γιατί δεν έχω πρόσβαση στις μελέτες. Και για να κάνω αυτή την αξιολόγηση χρειαζόμαστε περαιτέρω μελέτες. Είπατε πάνω από 800 μελέτες και μόνο κάποιες το αποδεικνύουν. Ποιες! Ποιο ήταν το μέγεθος των δειγμάτων, ποιες ήταν αυτές οι μελέτες. Το κρέας το μεταποιημένο είναι ένας παράγοντας ανεξάρτητος ο οποίος προκαλεί καρκίνο ή χρειάζεται να συντρέχουν και κάποιες άλλες περιστάσεις. Νομίζω ότι στην κατάσταση αυτή, μια που είναι τόσο σημαντικό το θέμα, έπρεπε να περιμένετε για τις μελέτες και να τις αναλύσετε πιο πολύ σε βάθος. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ. Και όντως είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η συζήτηση για ένα θέμα το οποίο έχει ευαισθητοποιήσει πολύ την κοινή γνώμη των ε, καταναλωτή, τον ανησυχεί του καταναλωτή. Ο κίνδυνος, παρότι είπατε ότι είναι παράγον πρόσληψης πρωτεϊνών ή ε, το κρέας και ότι δεν πρέπει βεβαίως και να ματαιωθεί τελείως ή να, να εκμηδενιστεί τελείως η καταναλωσή του, ασφαλώς μπορεί κάποιος καταναλωτής να αρχίσει να σκέφτεται ότι δεν πρέπει πια να καταναλώνει αλλαντικά ή κόκκινο κρέας και βέβαια ο παραγωγός μας, ο κτηνοτρόφος μας ε, ανησυχεί για τη συνέπεια στην κατανάλωση και την παραγωγή. Και επίσης μας λέτε ότι πρέπει να καταναλώνουμε τα φρούτα και λαχανικά. Ασ, ασφαλώς και το ξέραμε όλοι. Οι πιο πολλές είναι βεβαίως και το ξέραμε. Είναι παρόντα στα οποροκυπευτικά. Αλλά ξέρουμε ότι και αυτά έχουν και χημικά και ζυζανιοκτώνα και ούτω καθεξής. Ουσίες οι οποίες μπορούν να είναι καρκινογόνες με τη σειρά τους. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Μπορεί να αναπτύσσεται η παραγωγή των βιολογικών προϊόντων ολόχη αρκετά και όχι κατά τρόπο αρκετά λελογισμένο όπως θα λέγαμε, δηλαδή απλώς περιορίζεται η χρήση των ε, αλλά είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή για τον καταναλωτή, όπως επίσης ε, ξέρουμε ότι δεν συντηρούνται το ίδιο καλά ε, τα βιολογικά προϊόντα. Επίσης δεν μας μιλήσατε για το ψάρι. Ξέρουμε ότι το ψάρι, το καλό ψάρι που σέβεται και το περιβάλλον είναι καλό βέβαια για την κατανάλωση, είναι καλό για την υγεία, αλλά υπάρχουν και τα προϊόντα των ηχθειοτροφίων που επίσης γίνουν ανησυχίε. Και τα ψάρια που έχουν υψηλή ε, συγκέντρωση βαρέων μετάλλων ε, και ούτω καθεξής. Άρα ο κόσμος δεν ρωτάται τι να ταΐσει τα παιδιά του. Μήπως λοιπόν χρειάζεται μια πιο ευρεία και καθησυχαστική θα έλεγα για τον καταναλωτή ενημέρωση ώστε να αντιληφθεί ότι είναι η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων αλληλένδετε, ότι χρειάζονται προόδειες προς την ασφάλεια των, των τροφίμων, αλλά χρειάζεται ασφαλώς και πάνω απ' όλα πιο ευρεία ενημέρωση. Ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταλαβαίνετε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχει δημοσιεύσει την έκθεσή της αυτή η Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων ε, και το λέω ξεκινώντας ε, και δηλώνοντας ότι είμαι vegan εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή δεν τρώω κανένα προϊόν κρέατος ε, ζωικής προελεύσεως καλύτερα. Έχω δηλαδή στρατευτεί στο να μην καταναλώνω κανένα προϊόν ζωτικής προέλευσης εδώ και 20 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια βγήκαν κάποιες εκθέσεις στη δημοσιότητα που έδειχναν πόσο καταστροφικές για την υγεία μπορεί να είναι συνέπειες καταναλώσεις ε, κρέατος και γενικότερα περιέγραφαν ε, την αλλαγή, ε, μάλλον γενικότερα οδήγησαν σε μια αλλαγή στην κατανάλωση κρέατος, αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες γενικότερα στη Γερμανία έχει φτάσει στο 8% του γενικού πληθυσμού ο αριθμός των vegan, αυτών δηλαδή που δεν καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν, ε, και μάλιστα είναι αυξητικέ τάσει. Χωρίς όμως αυτό να έχει συνέπειες για τον παραγωγό ή τον κτηνοτρόφο, διότι βλέπουμε ότι έχει ανάπτυξη ο κλάδος αυτός διψήφια και είχα την ευκαιρία να συζητήσω στο 24ο ε, συνέδριο των παραγωγών κρεάτων στον Μπαντ Γκόντεσμπερκ πρόσφατα. Ε, συνομίλησα λοιπόν με τους παραγωγούς αυτούς, τους είπα ότι καλό θα είναι να κοιτάξουν να βρούνε και εναλλακτικές παραγωγές και μαθαίνω ότι σιγά σιγά και μάλιστα μεγάλη, πολύ μεγάλη όμιλη από τους μεγαλύτερους της Γερμανίας μετά τοπίζουν το επίκεντρο των ενδιαφέροντός τους και αντί για παραγωγή κρέατος αναζητούν εναλλακτικές, πράγμα το οποίο βρίσκω πολύ θετικό. Επίσης, για, το υψηλό, για την υψηλή περιεκτικότητα και σε λίπος, το 18% που λέμε κίνδυνο καρκινογένεσης, ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται και για μία αρρώστια της σύγχρονης εποχής ε, γιατί έχουμε τις υψηλές τιμές της ε, χολυστερόλης, ε, τα προβλήματα τα καρδιαγιακά και ενώ δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εναλλακτική η κατανάλωση ψαριών γιατί έχουν γίνει τόσο εντατικές αλλιεύσεις που ξέρουμε ότι σε δύο δεκαετίες δεν θα υπάρχει σε ελεύθερη βοσκή ε, ψάρια να καταναλώσει ο άνθρωπος. Τα δε, ηχθιο, ε, τα δε συστήματα ηχθειοκαλλιέργειας ε, είναι μάλλον πηγή αντιβιωτικών παρά άλλη τροφής, γιατί είναι γεμάτα με αντιβιωτικά τα ψάρια αυτά. Και βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με, τους, με, την ανθεκτικότητα των μικροβιών στα αντιβιωτικά. Άρα λοιπόν και φτάνω στο συμπερασμά μου. Έχουμε ...32 φορές περισσότερες εκπομπές τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το λέει μια άλλη έκθεση. Και αν θέλουμε να αντιστρέψουμε τις εξελίξεις κλιματικές αλλαγές... ...και να προστατεύσουμε τις μελλοντικέ γενιές... ...πρέπει να κάνουμε την κίνηση που απαιτεί η Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων, δηλαδή να παράγουμε και να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Είναι διαπιστωμένο ότι το τσιγάρο κάνει κακό στην υγεία του ανθρώπου και πάνω στο πακέτο των σιγαρέτων έχει επιβληθεί η αναγραφή ότι μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν και στις συσκευασίε ε, κρέατος να αναγράφεται ότι η υψηλή ή πολύ υψηλή κατανάλωση προϊόντος κρέατος μπορεί να θέτει τη ζωή μας σε κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χόσλιν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις εξηγήσεις που μας δώσατε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικές για να μπορούμε και να σχετικοποιούμε το όλο ζήτημα. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για κινδύνους που ε, μας απειλούν σε περίπτωση υψηλών καταναλώσεων κρέατος. Έχουμε δει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση να εκδηλώνεται σε παιδοκίνης γνώμης μέχρι ένα είδος αντιπαράθεσης πολιτιστικής θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι καλό να καταναλώνει κανείς βιολογικό κρέας βιολογικής προέλευσης κρέας σε χαμηλή ποσότητα παρά γενετικά τροπο, ε, τόφου από σόγια γενετικά τροποποιημένη. Τώρα, για την αναγραφή, αγαπητέ συνάδελφε, ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο και για την υγεία, είναι νομίζω υπερβολικό. Υπερβολικά υπερβολικό αυτό που προτείνατε. Αλλά θα ήθελα να δω εάν υπάρχει Φερρυπίν μια δυνατότητα να εκδοθεί, με το, ακολουθώντας το πράγμα της μια σύσταση να περιοριστεί η κατανάλωση του κρέατος. Πάνω απ' όλα πρέπει να σημειώσουμε ότι η υψηλή κατανάλωση κρέατος είναι αρνητική και το έχουμε δει γενικότερα. Το πρόβλημα είναι οι ποσότητες. Αυτό που καταναλώνουμε στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό ξεπερνά τα επίπεδα της λογικής και της υγείας. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια λογική και λογισμένη αντιπαράθεση ε, και συζήτηση για το τι παράγουμε, τι καταναλώνουμε, αλλά καλύτερα να μην αποδεθούμε σε μια πολιτιστική αντιπαράθεση η οποία θα σήμαινε ότι επιβάλλεται η θέση των βίγκανς ότι το κρέας πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία. Εν πάση ας μην προσπαθούμε να κάψουμε μαζί με τα ξερά και τα χλώρα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσίριο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παραδέχομαι ότι ανησυχώ όλος ιδιαίτερος. Ήλπιζα ότι ότι από τη συζήτηση αυτή θα καθισχαστούμε κάπως ή τουλάχιστον ε, θα είμαστε πιο ανακουφισμένοι. Ε, δεν αμφιβάλλω για την επιστημονική αξία των πορισμάτων αυτών και εγώ γνωρίζω από τέτοιου είδους μελέτες. Όμως ε, τέτοιου είδους εξέταση των θεμάτων αυτών από τον ΠΟΗ ουσιαστικά θα μπορούν να συνοδεύονται και από την κατάλληλη πολιτική επικοινωνίας. Διότι εάν εδώ αρχίσουμε να λέμε ότι αν ε, αρχίσω να τρώω πολύ κρέας, να πίνω πολύ καφέ, να καταναλώνω πολύ ζάχαρη, προφανώς μπορεί να κάνω κακό στο σώμα μου, στον οργανισμό μου. Αλλά στις μελέτες αυτές πρέπει να υποσημειώνεται ότι χρειάζεται και ένα σωστός τρόπο ζωής, ότι αν κάποιος είναι πιο νέος ή μεγαλύτερος ή αν έχει την τάδε την τάδε διατροφή, οι συνέπειες είναι διαφορετικές. Αν τα σοπεδώνουμε όλα και τα ε, μεταδίδουμε έτσι και στον τύπο και λέμε η μία ή η άλλη ουσία, το ένα το άλλο προϊόν ή τρόφιμο είναι καρκινογόνο όχι και θα ανακοινώνουμε, αυτό λες τα πάντα. Νομίζω ο οργανισμός αυτός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του αν τα δημοσιοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ προσπάθησα λοιπόν να το μελετήσω το θέμα και είδα ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που δημορφωνόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά διαβάζω ένα άρθρο του 2013 ενός από τα περιοδικά, τα περιοδικά για την ιατρική το Journal of Clinical Epidemiology ε, της, των ΗΠΑ που έκανε μια μελέτη η οποία σχετίζεται πλήρως με την τελευταία σύσταση του ΠΟΗ και ε, καταλήγει σε αποτελέσματα που είναι ανησυχητικά. Λέει ότι 55,5% των συστάσεών σας έχουν πολύ κακή επιστημονική τεκμηρίωση. Η δήλωση, η καταγγελία αυτή αυτού του περιοδικού τη εφημερίδα μάλλον, δεν την έκανε μια καθημερινή εφημερίδα την καταγγελία, αλλά ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίω. Ε, δεν είναι λίγο αυτό. Ε, ανησυχώ λοιπόν ιδιαίτερω για το πώ μεταδίδονται οι σχετικέ πληροφορίε. Εάν ε, οι πληροφορίε γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο, όχι απλώ ε, είναι εμπορικέ οι προτεραιότητέ μα, αλλά η προσέγγιση στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγάλο στοιχείο και τα επικοινωνικά σφάλματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Ένας οργανισμός που εκπροσωπεί ε, τα κάτι μέλη στον ΠΟΗ έχει κάνει μία δήλωση, έχει μάλλον εγκρίνει ένα ψήφισμα που ζητά ε, συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τις συστάσεις ε, των διαφόρων επιτροπών προκειμένου να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν αρκεί να πει κανεί ότι αν καταναλώσετε πολύ κρέας μπορεί να πάθετε καρκίνο ε, ή αν φάτε, καταναλώσετε πολύ ζάχαρη μπορείτε να πάθετε περισσότερο ή λιγότερο καρκίνο. Αυτό δεν αρκεί, αλλά αν συνεχίσουμε να δίνουμε τέτοιες πληροφορίες Πραγματικά δεν νομίζω ότι κάνουμε ιδιαίτερα πρόοδου. Ακόμη και στην ε, διατροφική εκπαίδευση του κοινού. Ε, υπάρχουν διαφορετικά διατροφικά προφίλ. Μια ιατρική μελέτη καθορίζει τελείως εν κενό το αν κάτι κάνει καλό ή όχι λες και ε, αρκεί μόνο για τροφή ή η κατανάλωση ε, ενός, άλλου προϊόντος για να είναι καλές καλά ή όχι. Όχι, χρειάζεται διατροφή, χρειάζεται σωματική άσκηση, χρειάζεται ένας καλός τρόπος ζωής. Αυτά λοιπόν είναι υπερπροστατευτικά και ε, νομίζω ότι πλήττουν την αξιοπιστία ενός τέτοιου έγκριτου οργανισμού όπως ο δικός σας, ο ΠΟΗ. Ευχαριστούμε και τώρα κυρίως Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι τις απόψεις όσων πήραν το λόγο και εξέφρασαν την επιφυλακτικότητά τους για την επικοινωνική πολιτική του ΠΟΗ. Ούτε και εμένα με έπεισε πολύ αυτή η προσέγγιση σα, βεβαίω. Χαίρομαι που η συζήτηση γίνεται, διότι είναι πραγματικά σημαντικό το θέμα. Εμεί από καιρό ακούμε διαφορετικέ απόψει επιστημόνων επανειλημμένος και μάλιστα αρκετά αξιόλογοι επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί σχετικά. Πολλά επιστημονικά λοιπόν στοιχεία είχαν ε, προλάβει τις δικές σας υποψίες και υπόνοιες. Βεβαίω, αν το κρέα και τα προϊόντα κρέατος καταναλώνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μπορεί να είναι καρκινογόνα. Ε, Συνήθω έχει κανεί 30% περισσότερο κίνδυνο. Εσεί λέτε κάτι διαφορετικό λιγάκι. 30% να παρουσιάσει διαφορετικά είδη όγκων, όχι μόνο του ορθού, αλλά του παγκρέατος, της σχολή, των πνευμόνων και το καθεξής. του σηκωτιού, του ύπατος και το καθεξής. Όλα αυτά σχετίζονται με τις λειτουργίες του μεταβολισμού. Ε, αυτά λοιπόν έχουν ήδη υποθεί στο παρελθόν. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Και αν διαβάσω αυτό που μόλις είπε ο συνάδελφός μου, αν διαβάσω ότι λέτε στην ανακοίνωσή σα και για τα επιστημονικά θεμέλια των πορισμάτων σα, <clears throat> για μένα δεν καθίσταται σαφέ το εξή. Ε, φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα θέλουμε να το κενώσουμε και από κάθε ουσία. Ε, λέμε ότι το 18% αύξηση κινδύνου για τον καρκίνο του ορθού ε, αφορά τα προϊόντα κρέατος και τα κόκκινα κρέατα μήπως έπρεπε να, να παραμείνουμε μόνο στο κρέας διότι το σύνολο των δεδομένων έχει μεταδοθεί και συνδυαστεί και με άλλα γνωστά στοιχεία που ήταν γνωστά και από την επιστημονική βιβλιογραφία. Επίσης, γιατί τι έκθεση μιλάμε στους παράγοντε κινδύνου, γιατί και αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Δεν μπορώ να λέμε αυξάνεται κατά 18% κίνδυνος χωρίς να αναλόγως να ορίζουμε και την, το ποσοστό έκθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λίγο πολύ, είναι όλα σχετικά. 18% είναι μια απόλυτη δήλωση, ένας απόλυτος αριθμό. Είναι λοιπόν ε, σαφές, ε, σημαντικό να γνωρίζουμε πόση τέτοια ποσότητα πρέπει να καταναλώσω για να παρουσιάσω 18% πιθανότητας άξισης. Ε, επίσης για τις εκτιμήσεις. Ε, τα συγκρίνατε με τον συνδυασμένο κίνδυνο, όπως είπε προηγουμένω και μια άλλη συνάδελφος, με τον συνδυασμένο κίνδυνο άλλων ε, επικίνδυνων παραγόντων. Διότι πάλι είναι όλα σχετικά. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε τον κίνδυνο σε εργαστηριακές συνθήκες ε, και να το συγκρίνουμε με τον κάπνισμα και το αλκοόλ χωρίς να σκεφτόμαστε τον συνδυασμό που μπορεί να παρουσιάσουν τα επικίνδυνα στοιχεία. Αυτό και, και... και αυτό μάλλον είναι πολύ σημαντικό για να ξορκίσουμε έναν φόβο τον οποίο βρίσκω πολύ βάσιμο. Δηλαδή, η βιομηχανία τροφίμων που έχει πολύ μεγάλες ε, δυνάμεις, είναι πολύ ισχυρή, ήθελε κάπως να κενώσει το νήματό τη στην ε, ανακοίνωσή σας, στην μελέτη αυτή. Βεβαίως, γιατί υπάρχει και μέλημα για την, ε, μια μέρημνα για την υγεία, αλλά και για τα οικονομικά της συμφέροντα. Από την επιστημονική όμως σκοπιά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, να ε, διευρυνθεί το πεδίο της μελέτης, το είδος της αξιολόγησης και εκτίμησης πρέπει να γίνει και να υιοθετηθεί μια επιστημονική μεθοδολογία αυτόνομη και ανεξάρτητη για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο ε, γίνεται πιο κοντινό στην πραγματικότητα και να, και εμείς, να μπορέσουμε και εμείς να ρυθμίσουμε τις μελλοντικές μας συμπεριφορές αναλόγως. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως καταλαβαίνω ποια είναι η θέση του ομιλητή. Είναι υποχρεωμένος λόγω της θέσης του. Βασιζόμενος στα στοιχεία τα οποία έχουν φτάσει στα μάτια του να μας πει πως το κόκκινο κρέας είναι καρκινογόνο. Εάν όντως υπάρχει σχετικό έβριμα στις μελέτες. Όμως αυτή η δήλωση είναι παραπλανητική γιατί αυτό το 18% που δίνεται και που είναι ενδεικτικό του κινδύνου θα πρέπει να συγκριθεί με τον κίνδυνο του καπνίσματος για παράδειγμα που ήμασταν στο 2.500%. Αλλά για τον απλό άνθρωπο αυτό το 18% τι σημαίνει ότι ένας στους 6 θα νοσήσουν. Και αυτό είναι παρανόηση, είναι παραπλάνηση. 18% σε ποιο στο εφαρμόζεται. Επίσης, παρατηρήσατε πως υπάρχει και ένα παράδειγμα του τι θα συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η κατανάλωση κρέατος είναι κυρίως μεταποιημένου ε, ή προπαρασκευασμένου κρέατος. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε κατανάλωση νοπού κρέατος. Εκεί μειώνεται ο κίνδυνος. Επίσης προκύπτει το εξή ερώτημα. Οι περισσότερε από αυτέ τι μελέτες έχουν γίνει ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου υπάρχει κλωνοποιημένο κρέας που κυκλοφορεί στην αγορά. Ε, κρέας που έχει περάσει από ακτινοβολία για να συντηρηθεί. Νομίζω λοιπόν πως αν αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε ευρήματα από τη ΣΥΠΑ, ενδεχομένως να μας παραπλανούν. Τώρα, αν πιστεύουμε πως ο κίνδυνος αυτός είναι σοβαρός, τότε πριν από δύο εβδομάδες πήραμε τη λάθος απόφαση στο Στρασβούργο όταν αφαιρέσαμε τις επιδοτήσεις από τις σταυρομαχίες γιατί τελικά αν δεν επιτρέπεται η κατανάλωση του κράτους μήπως θα έπρεπε μόνο τις σταυρομαχίες να στηρίζουμε. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ λέει κυρία Ντογνανού, δεν θα σας κουράσω. Με ανησυχεί ιδιαίτερα σε αυτή η ε, έκθεση για τα κόκκινα κρέατα, για τα κατεργασμένα και με προβληματίζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί όπως είπε η κυρία Γροστέτ, και οι εντατικές υδατοκαλλιέργειες ε, και το ψάρια που προέρχεται από αυτές ή τα απορρολαχανικά που έχουν καλλιεργηθεί με τη χρήση των σανιοκτώνων, πιστεύω, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίστοιχα πορίσματα σε μια τέτοια έκθεση. Ε, θα βρίσκατε κάτι δηλαδή να πείτε. Ρωτώ λοιπόν εάν υπάρχουν γενετικές προδιαθέσεις οι οποίες να μπορούν να δείξουν μια ευαισθησία στην κατανάλωση ε, κόκκινου κρέατος, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, έχετε κάνει διαφοροποίηση ε, ζώα που έχουν εκτραφεί με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ενδεχομένως περισσότερους καρκίνους. Ε, τρίτον, υπάρχει διαφορά σε σχέση με την κατανάλωση βιολογικής προελεύσεως κρέατος και βιομηχανικής παραγωγής. Και για την σήμανση, γιατί βλέπω κάτι το υποκρουστικό εδώ. Μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία δημοσιεύει ε, μια ετικέτα η οποία δείχνει μια μπριζόλα με το κόκαλο για το μπάρμπεκιου και από κάτω η ετικέτα γράφει «Αλιευθέν στον Ατλαντικό» για να καταλάβουμε πόσο αξιόπιστες είναι οι ετικέτες στα σούπερ μάρκετ. Ε, κυρία Εύη, ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω πολύ τον εκπρόσωπο του ΠΟΕ για την παρουσίασή του, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι τα πάντα τα ε, ισοπεδώνουμε και τα οδηγούμε σε μια απλή επιστημονική εξήγηση. Όταν είναι αρεστά ε, τα στοιχεία που ανακοινώνονται, οι αντιδράσεις είναι θετικές και αντιστρόφως. Εγώ χαίρομαι για την παρουσίαση αυτή. Προσωπικά είμαι φυτοφάγος κατά το ίμιση της διάρκειας της ζωής μου και είμαι πεπισμένη ότι έχουμε πολλές προσωπικές επιλογές να κάνουμε για την ε, κατανάλωση και τη διατροφή μας και θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να έχουμε και ειδικότερες πιο συγκεκριμένε συστάσεις από την πλευρά των πολιτικών ευθυνόντων. Επ' αυτού πιστεύω ότι η έκθεση μπορεί να δώσει την αφορμή για μια ε, εντελεχή μελέτη του όλου θέματος. Διότι δυστυχώς πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε για την ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση, την υπερβολική κατανάλωση κρέατο, υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο θέμα που ε, εγείρει η όλη μελέτη. Το θέμα της εντατικής εκτροφής και κτηνοτροφίας και εντατικής παραγωγής κρέατος που συζητήσαμε μόλις σήμερα. Ε, πόσο επηρεάζει η εντατική παραγωγή τις κλιματικές αλλαγές, την απώλεια πόρων, την ε, διασπάθηση των πόρων, την αποψήλωση, την απερίμωση και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το τεράστιο θέμα. Όλα αυτά είναι λέμβετα. Όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Πρέπει να έχουμε περισσότερο συνειδητέ επιλογές για το μέλλον μας, διότι η κατανάλωση και η παραγωγή κρέατος ως τώρα μας οδηγεί στην ε, υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων μας, που ο πλανήτης μας δεν την αντέχει άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα δικά σας τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε πόη. Δεν νομίζω πως σε αυτή τη φάση έχω πολλά να προσθέσω. Εμείς σίγουρα καταγράψαμε τα σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση και αναμένουμε ε, την δημοσίευση της ε, μελέτης που θα απαντήσουν ε, κάποια από τα ερωτήματα που θέσαμε. Όπως είπε και ο κύριος Μπερτολίνη, το θέμα με τα κρέατα και τον καρκίνο κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τώρα από τη σκοπιά της ε, Κομισιόν και για να δούμε την ε, δημόσια υγεία και το βάρος που είναι τα χρόνια, οι χρονίες παθής και ο καρκίνος για την Ευρώπη, προφανώς η άσκηση και οι καλές διατροφικές συνήθειες ε, πάνε χέρι-χέρι και θα πρέπει να εξετάζονται πάντα. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι η ορθότερη τακτική. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Σίγουρα ανησυχούμε ιδιαίτερα για το πώς ε, εξαπλώνεται ο καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρους ε, ένας από αυτούς που μας απασχολεί περισσότερο με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προληπτικές εξετάσεις. Το εξετάζουμε λοιπόν με προσοχή, παρακολουθούμε τις λεπτομέρειες, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, στις επιστημονικές μελέτες και με χαρά θα διαβάσουμε τη μελέτη μόλις δημοσιευθεί σε κάποιους μήνες. Ευχαριστώ. Thank you very much. now... Ευχαριστώ. Ύστερα από αυτή την έντονη συζήτηση θέλουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και γιατί ήταν πολύ έντονη η αντιπαράθεση στις εφημερίδες τελευταία εβδομάδα. αλλά και γιατί νομίζω ήταν πολύ σαφής και συνέπειες για την αγορά κρέατος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση και να πούμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αλλά και τις συνθήκες μας τις οποίες έχουν εκπονηθεί οι, συνθ... οι μελέτες. Γιατί υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι, μας είναι γνωστά για να παίρνουμε αποφάσεις. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές που έλαβαν ε, το λόγο και έκαναν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Ξεκινώ με ένα πρώτο σχόλιο, το οποίο κρίνω πολύ σημαντικό και θα ήθελα να πω ότι είναι και το ζήτημα η ε, το οποίο πεσήμαναν ορισμένοι από εσά, δηλαδή η καθυστερημένη δημοσίευση της έκθεσης. Συμφωνώ, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε και εμάς εσωτερικά. Η πλήρης έκθεση, η οποία καταγράφει συνοπτικά όλες τις μελέτες και τις λεπτομέρειες ε, της βιβλιογραφίας κτλ, είναι υπό αναθεώρηση και επανεξέταση έτσι ώστε όλες οι παραπομπές μας και όλα τα άρθρα που έχουμε αξιοποιήσει να επαληθευθούν ε, προσεκτικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα απορίσματα γιατί η ανάλυση έχει γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν πρόκειται να αλλάξει τα αποτελέσματα. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι θα, πρέπει να γίνεται, θα έπρεπε να γίνεται ταυτόχρονα δημοσίευση. Ε, προσπαθούμε να το αποφύγουμε για το μέλλον και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Κάποια σχόλια που είχαν να κάνουν με τις διατροφικές συνήθειες, την καταναλώση κρέατος και τις συνέπειες στην υγεία. Είτε λόγω επιμόλυνσης σε φυτικά προϊόντα, είτε για άλλους ε, λόγους. Νομίζω ότι είναι τμήμα μιας άλλης συζήτησης για την υγιεινή διατροφή που πρέπει να γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο και πρέπει να συζητηθεί πιστεύω και εδώ το ζήτημα της ε, επιβάρυνσης της υγείας από τα αλκοολούχα, από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης κτλ. Αλλά είναι άλλη συζήτηση, όπως είπα, αυτό που σας παρουσιάζουμε εδώ και παρουσιάζουμε στην, και στην επιστημονική κοινότητα, όπως και στην ευρύτερη κοινή γνώμη, είναι απαντήσει στο ερώτημα ως προς την καρκινογενετικότητα του κρέατος ε, νοπού και κατεργασμένου. Αυτή είναι η απάντηση και βεβαίως την εγγράφουμε στο ε, πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής όπου μπορούμε να πούμε ποιος, πως μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι αποδεκτή. Έχουμε πει πιστεύω επανελειμμένως και στις συστάσεις μας για την υγιεινή διατροφή ότι αυτό ισχύει. Δεν αντικρούονται ε, από αυτό γεγονός τα ε, πορίσματα της έκθεσης, οι επιστημονικές ε, αναλύσεις, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίριο, ε, είναι ακριβής. Ξέρω τη μελέτη στην οποία αναφερθήκατε και αυτή έχει υποστεί πολλές επικρίσεις εσωτερικά αλλά και από άλλους ερευνητέ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συστάσεις της ΠΟΗ μπορεί να αποτελούν πηγή ερωτηματικών γιατί θεωρείται ότι δεν είναι η επιστημονική βάση γερή όπως θα όφιλε αυτό ιδίω στο παρελθόν βέβαια συνέβαινε, αλλά πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή από εδώ και μπρο, οτιδήποτε δημοσιεύεται, οτιδήποτε κείμενο εκδοθεί από την ΠΟΗ έχει περάσει μέσα από τέτοιο ξεσκόνισμα και έρευνα και αναθεώρηση που πολλέ φορέ αναγκαζόμαστε να πούμε φτάνει, μην προχωρήσετε, μην κάνετε κι άλλη ανάλυση γιατί ε, θέλουμε να είμαστε στο δυνατόν πιο ακριβείς και ασφαλείς ω προ τι συστάσει μα. Μπορεί στο απότερο παρελθόν να συνέβαινε αυτό, γιατί εγώ στο δεκαετία του 70 δεν ήμουν στην ε, ΠΟΗ δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά αυτό που λέτε δεν ισχύει. Και ξέρω για τη μελέτη του 2013 που αναφέρατε, που υπέστη, ή το υποβλήθη και μάλλον σε πολλές επικρίσεις λόγω ακριβώς κάποιων ασαφών διασύνδεσεων με κάποιους τομείς. Για το κόκκινο κρέας, πω και κατεργασμένο και ο κίνδυνος κατανάλωσης 100 γραμμαρίων σε σχέση με την μη κατανάλωση κόκκινου κρέατος ε, είναι 17% όχι 18% που ακούστηκε για το κόκκινο κρέας και 18% για το ε, κατεργασμένο κρέας σε ποσότητες 100 γραμμάρια για τον οπό κρέας και 50 γραμμάρια για το κατεργασμένο κρέας και σε σχέση με το να μην καταναλώνεται καθόλου κρέας. Σε αυτό που αναφέρθηκε η ε, αλληλεπίδραση διαφορών παραγόντων. Φυσικά και κάποιος ο οποίος καπνίζει αλλά ταυτόχρονα εκτίθεται και σε αμίαντο έχει πιο πολύ πιθανότητα να πάθει καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με κάποιον που δεν καπνίζει ή δεν εκτίθεται σε αμίαντο. Ε, αυτό που λέμε εμείς για τον κίνδυνο καρκίνο του ορθού είναι ακριβώς η συγκεκριμένη αναζήτηση της καρκινογενετικότητας του κρέατος κόκκινου κρέατος στις διάφορες εκδοχές του. Αλλά ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων περιβαλλοντικών ή λοιπόν. Αναφέρεται επίσης ότι χρειάζεται ανεξάρτητη έρευνα. Και για να είμαι ειλικρινής, είμαι επιφυλακτικός ως προς την δήλωση αυτή, γιατί η έρευνα που σας παρουσιάζουμε είναι η πλέον ανεξάρτητη που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Με επιστήμονες, με 100 τουλάχιστον δημοσιεύσεις από επιστημονικά ε, περιοδικά και επιθεωρήσεις επιστημονικές που ε, εκλήθησαν να αναθεωρήσουν και μάλιστα κλεισμένοι επί δέκα μέρες μέσα σε μια αίθουσα για να μην έχουν καμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Πιο ανεξάρτητη έκθεση από τη δικιά μας δεν μπορεί να γίνει εκτός και να έχετε να μας προτείνετε εσείς κάτι και πολλές φορές να τα ακούσουμε για τον τρόπο και το στυλ της εκθέσεως. Κοιτάξτε, οι μελέτες έχουν αναλυθεί και πρέπει ιδιαίτερα να πω ότι δόθηκε έμφαση σε μελέτες που όριζαν μια πληθυσμιακή ομάδα και την παρακολουθούσαν για 20-30 χρόνια. Πληθυσμιακές εκθέσεις που έχουν γίνει και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η μελέτη EPIC, πολύ σημαντικές μελέτες και έρευνες που παρακολουθούν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες σε διάφορες χώρες ευρωπαϊκές και όχι μόνο τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι λοιπόν μια γενική επισκόπηση των συνεπειών της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και θέλω να σας υπενθυμίσω τον βιολογικό μηχανισμό που δεν έχει να κάνει με την προέλευση του κρέατος του, αν είναι δηλαδή ε, βιολογικής παραγωγής με, ε, εκτροφή με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κλπ. Έχει να κάνει με τη μοριακή σύσταση του κρέατος και τον τρόπο της του ψησίματος του. Δεν σας λέω ότι είναι καλύτερα φάτε βιομηχανικό και παραγωγής ε, προϊόν ε, σε σχέση με το βιολογικό το οποίο προέρχεται από ένα πολύ καθαρό περιβάλλον κλπ. Βεβαίως πάντα θα είναι καλύτερο το δεύτερο. Αλλά στη μελέτη μας ε, η εστίαση ήταν στην βιολογική σύσταση του κρέατος, στην, βιολογική, στην μοριακή συμπεριφορά του κρέατος. τα συμπεράσματα. Όντως, θα συμφωνήσω μαζί σας, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα επικοινωνιακό. Είναι το σωστό αυτό και γι' αυτό έρχομαι να μιλήσω εκ μέρου του Γενικού Διευθυντή μα του Δόκτωρ Τσάνγκ, που με παρακάλεσε να έρθω να σας μιλήσω. Έχει γίνει εσωτερική συζήτηση και διάλογο. Θα, αναλύσουμε και πάλι τα ζητήματα αυτά και σα ενημερώνω ότι θα γίνει ανα, ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών και από άλλο πάνελ πολύ σύντομα ε, πάνελ το οποίο θα τα εξετάσει και υπό το πρίσμα μιας υγιεινής διατροφής ώστε να προτείνουμε στο ευρύ κοινό ποσότητες που θα μπορούσαν να είναι μια λογική ημερήσια πρόσληψη. Αυτά στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής που είναι πολύ σημαντικό επίσης. Κύριε Λαβία, δεν νομίζω να έχω τίποτα άλλο να προσθέσω και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για τα όσα μας είπατε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κάτι ξέχασα, ναι. Για την κατανάλωση στην Ευρώπη. Να σας πω πως έχουμε στοιχεία από μία μελέτη, μελέτη EPIC, δηλαδή μεταποιημένα κρέατα, το μέσο, Ελλάδα, 11 με 19 γραμμάρια την ημέρα, και αυτό είναι το χαμηλότερο, και στην Νορβηγία είναι 48 την ημέρα για τις γυναίκες και 95 στη Γερμανία για τους άνδρες την ημέρα. Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία γιατί κάποιος μου ζήτησε, με ρώτησε την ψαλίδα ε, για το που βρίσκεται η κατανάλωση. Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με τη συζήτηση αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, ε, εύκολο το καθήκον σας σήμερα. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε το απόγευμα στις 3.